So, dear colleagues, ladies and gentlemen. Λοιπόν, συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, παρακαλώ καθίστε, το πρόγραμμα μας είναι πιεσμένο. Of first like to Βεβαίως, πρώτα απ' όλα να καλωσορίσω τον υποψήφιο Επίτροπο Εμπορίου, τον κύριο Χόγκαν που κάθεται εδώ. στόχος ε, της συνεδρίας είναι προφανής. Ο ε, κύριος ε, Χόγκαν έχει απαντήσει στις γραπτέ ερωτήσεις, τις οποίες έχετε λάβει και έχουν δημοσιευτεί και στην σελίδα του Κοινοβουλίου. Και να σας ενημερώσω επίσης πως η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων δεν έχει κάποια αντίρρηση για τη διεξαγωγή της σημερινή ακρόασης, οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε κανονικά. Και ναι, Κύριε Χόγκαν, καλώς ήρθατε και πάλι στην Επιτροπή μας. Την δημοκρατική καρδιά της εμπορική πολιτικής. Βεβαίως είναι μεγάλη τιμή για μένα να προεδρεύω και όπως και η εμπορική πολιτική έχει πραγματικά εξελιχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Τώρα η Επιτροπή μας είναι η Επιτροπή εκεί είναι η οποία εγκρίνει ή όχι τις εμπορικές συμφωνίες και επίσης ε, εμπλέκεται και στην σχετική νομοθεσία. Είναι λοιπόν η δημοκρατική φωνή των πολιτών της Ευρώπης στην εμπορική πολιτική. Και ναι, ζούμε σε καιρούς δύσκολους. Η σχέση μας με τους εταίρους μας ε, είναι περίεργες για διάφορους ε, λόγους. Πιθανώς θα έχουμε Brexit ε, προσεχώς και από μέρα σε μέρα θα έχουμε και δασμούς από τις ΕΠΑ με βάση την απόφαση του ΠΟΕ για την Boeing. Ευτυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταφέρει να ε, διαπραγματευτεί καλές διμερείς ε, εμπορικές συμφωνίες ε, και καλές εμπορικές σχέσεις για να σταθεροποιήσουμε το παγκόσμιο σύστημα εμπορίου. Και βεβαίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει παίξει έναν σημαντικό ρόλο στην ε, βελτίωση των εμπορικών συμφωνιών όπως κάναμε στην ΣΥΤΑ. Στην ομοθεσία όπως κάναμε παραδείγματος χάρη για τα ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων και ναι, το εμπόριο βεβαίως είναι κάτι το οποίο απασχολεί την ε, κοινή γνώμη. Ο κόσμος, ε, η κοινή γνώμη θέλει να γνωρίζει ποιος ωφελείται, εάν το εμπόριο εξασθενίζει την προστασία των καταναλωτών και κατά πόσον συνεισφέρει στην ε, Συμφωνία των Παρισίων. Αρκετές προκλήσεις λοιπόν, όμως θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε και να πάρουμε στα σοβαρά την εμπορική πολιτική με βάση κάποιες αρχές. Η βιωσιμότητα θα πρέπει να είναι μία από αυτές. Το εμπόριο ως αποτελεσματικό εργαλείο για δίκαιες προδιαγραφές για τα αγαθά και βεβαίως για την διαδικασία παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών και βεβαίως και οι συμβάσεις του ILO παίζουν σημαντικό ρόλο. Δεύτερον, εφαρμογή και επιβολή. Για εμένα είναι σαφές ότι έχει φτάσει η στιγμή να περάσουμε από τα λόγια στις ε, πράξεις. Το ευρύ δίκτυο εμπορικών ε, συμφωνιών που έχουμε θα πρέπει να έχει αποτελέσματα εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρειαζόμαστε τα απαραίτητα μέσα γι' αυτό. Τρίτον, συνοχή. Η εμπορική πολιτική θα πρέπει να είναι συνεκτική με τις άλλες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο εθνικό επίπεδο. Παραδείγματο χάρη δεν έχει νόημα να ζητάμε μείωση των επιδοτήσεων στην αλία και ταυτόχρονα προσπαθούμε να επιδοτήσουμε νέα αλληλευτικά σκάφη. Πρέπει να είμαστε λοιπόν συνεπείς στην πολιτική μας και επίσης ε, μια πολιτική η οποία θα ανταποκρίνεται στον δημοκρατικό έλεγχο. Η Ούρσουλα Φοντερ Λάιν έχει πει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ειδική σχέση μεταξύ Κομισιόν και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και κύριε Χόγκαν, αφού διάβασα τις γραπτές σας απαντήσεις, νομίζετε αυτήν την θέση. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ σε τέσσερα σημεία στα οποία θα θέλαμε περισσότερες διευκρινήσεις. Πρώτα απ' όλα, ε, είμαι πεπισμένος ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να θεωρείται ως ένα ε, θεσμικός δρόν μετά τις εξελίξεις των τελευταίων ε, δέκα ετών και να μην θεωρείται απλώς ε, ένα ενδιαφέρον μέρος στις απαντήσεις 3 και 7 δεύτερον. Βεβαίως υπάρχει δέσμευση για να μοιραστείτε τα έγγραφα διαβούλευσης, κάτι το οποίο είναι μια βελτίωση της υφιστάμενης ε, κατάστασης, αλλά κύριε Χόγκαν, ίσως ε, κάτι τέτοιο δεν αρκεί. Αυτά συντάσσονται με τα κράτη-μέλη και είναι σαφές ότι η σημαντική ε, εργασία γίνεται πριν συνταχθούν αυτά τα έγγραφα. Οπότε οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώνονται με τα έγγραφα αυτά, οπότε εμείς θα θέλαμε ενημέρωση πριν ολοκληρωθούν αυτά τα έγγραφα. Τρίτον, ταυτόχρονα, θα ήθελα να έχουμε μεγαλύτερες έπαφες στο θέμα της προσωρινής εφαρμογής η Ursula von der είπε ότι η Κομισιόν θα πρέπει να προτείνει προσωρινή εφαρμογή μόνο αφού έχει δώσει τη σύμφωνη γνώμη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η δική σας απάντηση δεν ήταν τόσο σαφής και θα ήθελα να επανέλθετε σε αυτήν και να ξεκαθαρίσετε ότι τα δημοκρατικά δικαιώματα του Κοινοβουλίου θα γίνουν σεβαστά στο θέμα αυτό της ε, προσωρινής εφαρμογής. Και τέταρτον, η, εξέταση, ε, η αρμοδιότητα εξέταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να αφορά και την εφαρμογή υφιστάμενων συμφωνιών. Εμείς ως Επιτροπή είμαστε σαφείς ότι οι μικτές επιτροπές, ε, τα συμβούλια και οι άλλοι οργανισμοί που μπλέκονται στην ε, εφαρμογή των συμφωνιών δεν θα πρέπει να είναι μαύρα κουτιά, θα πρέπει και αυτά να δέχονται τον δημοκρατικό έλεγχο. Κυρίε και κύριοι. Πρόκειται για μια καθοριστική στιγμή του κοινοβουλευτικού ελέγχου της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως θα ζητήσω από τους συναδέλφους μου να εκφράσουν την απόψή τους με σαφείς ερωτήσεις, με τον σαφή στόχο να αποσπάσουν σαφείς δεσμεύσεις από εσάς, τον νέο Επίτροπο. Ε, δεν πρόκειται λοιπόν απλά για μία ανάκριση. Πρέπει να αποτελέσει ένα σημείο καθορισμού της κοινή στρατηγικής μας για την εμπορική πολιτική τα επόμενα πέντε χρόνια. Οπότε, περνάω τώρα στα πρακτικά. Πρώτα απ' όλα, η δομή της ακρόασης πρέπει να ακολουθήσει βεβαίως όλο τον κανονισμό του Κοινοβουλίου και θα πρέπει να δοθεί μια δίκαιη και η ευκαιρία σε όλους τους υποψήφιους επιτρόπους να παρουσιάσουν εαυτούς και τις απόψεις τους. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν, ο κύριος Χόγκαν έχει την δυνατότητα να κάνει μια αρχική δήλωση 15 λεπτών. Και μετά, σύμφωνα με τον κανονισμό, θα έχουμε χρόνο για 25 ερωτήσεις από τους βουλευτές. Στο πρώτο μπλοκ ερωτήσεων θα έχουμε τις ερωτήσεις των 7 συντονιστών των πολιτικών ομάδων στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και στο δεύτερο γύρο θα έχουμε ερωτήσεις από 18 βουλευτές σύμφωνα με την ποσόστοση που δίνεται στην κάθε πολιτική ομάδα περιλαμβάνοντας και εκπρόσωπο των μη εγγεγραμμένων βουλευτών. Και Καλωσορίζω αυτή τη στιγμή τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών, τον κύριο Ντέιβιντ Μακάλιστερ, ο οποίος ε, και αυτός θα κάνει ερωτήσεις μαζί με τους 18 βουλευτές. Οι ερωτήσεις και απαντήσεις θα γίνουν σε διαστήματα των 5 λεπτών. Ο κάθε βουλευτής λοιπόν έχει ένα λεπτό για να κάνει την ερώτησή της. Μετά Κύριο Χόγκαν έχει την ευκαιρία να δώσει μια δίλεπτη απάντηση και μετά, εάν απαιτηθεί, υπάρχει δυνατότητα για τον ίδιο ή την ίδια βουλευτή να κάνει μια ερώτηση ε, ακόμα maximum ενός λεπτού. Και πάλι ο υποψήφιος επίτροπος έχει τη δυνατότητα να απαντήσει σε ένα λεπτό. Είναι σαφής νομίζω οι κανόνες ότι η δεύτερη ερώτηση πρέπει να αφορά την απάντηση στην πρώτη ερώτηση και να μην αφορά άσχετο ζήτημα. Οπότε φυλάσσομαι του δικαιώματος να μην επιτρέψω μια δεύτερη ερώτηση εάν δεν ανταποκρίνεται σε αυτό το κριτήριο. Και έτσι θα διεξαχθεί η συζήτηση. Στο τέλος των ερωτήσεων, ο, Επιτροπός, ε, ο υποψήφιος Επιτροπός θα έχει άλλα πέντε λεπτά να κάνει μια ε, δήλωση για να ολοκληρώσει. Όπως σας είπα, ο χρόνος μας είναι αυστηρά περιορισμένος στις 3 ώρες. Άρα είναι αυστηρά περιορισμένος και ο χρόνος για να γίνουν ερωτήσεις και θα επιβάλλω τα χρονικά όρια. Η διερμηνία παρέχεται και στις 23 γλώσσες και βεβαίως σε αυτήν την ε, συνεδρία, σε μια που έχουμε τον Ιρλανδό ε, Επίτροπο και έχουμε και Ιρλανδούς βουλευτές, μπορούν να μιλήσουν και την γλώσσα τους. Όλοι οι βουλευτές μπορούν να μιλήσουν την μητρική τους. Θα ήθελα όμως να σας υπενθυμίσω ότι θα πρέπει να παραμείνετε εντός του χρόνου. Και λόγω του ότι έχουμε ακριβώς ε, διερμηνία, να σας παρακαλέσω να μιλάτε κάθαρα και όχι πολύ γρήγορα για να μεταφραστείτε και βεβαίω να φανεί και προς τα έξω γιατί ω συνήθω η συνεδρίαση της Επιτροπής μας μεταδίδεται ζωντανά στην σελίδα του Κοινοβουλίου και καταγράφεται. Αυτά ως εισαγωγή για το πώς θα διεξαχθεί αυτή η διερμηνία και τώρα θα ζητήσω από τον υποψήφιο Επίτροπο Εμπορίου, τον κύριο Χόγκαν, να κάνει την αρχική του τοποθέτηση. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές. Είμαι ιδιαίτερο ευγνώμων στην υποψήφια πρόεδρο τη Κομισιόν, την κυρία Φοντερ που με όρισε επίτροπο αρμόδιο για θέματα εμπορίου και ελπίζω ότι στο τέλο τη ακρόαση αυτή θα θεωρήσετε ότι μπορείτε να μου εμπιστευτείτε το ρόλο αυτό. Άλλωστε το διεθνέ εμπόριο δεν μου είναι άγνωστο. Ω αρμόδιο για την Γεωργία Επίτροπος ε, συνεργάστηκα στενά με την απερχόμενη Επίτροπο Σεσίλια Μάλστρομ η οποία αφήνει πολύ θετική κληρονομιά πίσω τη και ελπίζω να οικοδομήσω πάνω σε αυτή την κληρονομιά. Επίσης από πρώτο χέρι έχω δει πόσο ζωτικό ρόλο έχει το διεθνές εμπόριο για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία στις 7 θέσεις εργασίας έχουν να κάνουν με την εξαγωγή αγαθών και υπηρεσιών. Πιστεύω λοιπόν ότι η εμπορική πολιτική της Ένωσης μπορεί και πρέπει να παρέχει πραγματικές δυνατότητες για βιώσιμη ανάπτυξη, σταθερότητα και προβλεψιμότητα σε έναν όλο και πιο ρευστό κόσμο. Ταυτόχρονα προσφέροντας ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις της Ένωσης και προστασία από αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Όμως η εμπορική πολιτική πρέπει να μπορεί και να εξελίσσει Πρέπει να μπορούμε να καταδείξουμε ότι μπορεί να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις για την ασφάλεια, για τη στρατηγική αυτονομία και την τεχνολογική ηγεσία. Επίσης, να αντικατοπτρίζει και να προωθεί τις αξίες μας, το τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, στον τομέα της κλιματικής δράσης, της βιώσιμης ανάπτυξης, των εργασιακών δικαιωμάτων, ε, τα πρότυπα, την ε, ενδυνάμωση και χειραφέτηση των γυναικών. Πριν ε, περάσω στις προτεραιότητές μου, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω πως εφόσον εκλεγώ θα συνεχίσω να εργάζομαι με διαφανή τρόπο, όπως ε, άλλωστε στο τελευταίο κοινοβούλιο η εμπορική πολιτική χαρακτηριζόταν από αυτή τη διαφάνεια. Θα έρχομαι τακτικά στην Επιτροπή σας, καθώς και στην Ολομέλεια ε, και επίσης ε, θα σας παραχωρώ έγκαιρη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που θέλετε. Θα λάβω πολύ σοβαρή υπόψη αυτά που είπατε κύριε Πρόεδρε. Επίσης θα παροτρύνω το Συμβουλίο να ακούει τις απόψεις σας για να σημειωθεί η πρόοδος σε νομοθετικά ζητήματα και βέβαια να έχετε εσεί πρώτα τη δυνατότητα να δίνετε σύμφωνη γνώμη σας πρώτα εφαρμοστούν εμπορικέ συμφωνίε. Θα συνεργαστώ μαζί σα ε, για να εξηγήσουμε, προωθήσουμε τον την εμπορική μα πολιτική. Ε, χρειάζεται να υπάρχει ακριβή επαγγελματική επικοινωνία ε, και ενημέρωση για τι εμπορικέ σχέσει. Έρχομαι λοιπόν τώρα στι πέντε βασικέ μα προτεραιότητες. Πρώτα απ' όλα πρέπει να στηρίξουμε σταθερή, προβλέψιμο ε, εμπορικό περιβάλλον βασισμένο σε κανόνε, ενδυναμώντα τον ΠΟΕ, τον Οργανισμό με εμπόριο. Ταυτόχρονα πρέπει να διαχειριστούμε τις βασικές αυτές σχέσεις που έχουμε και να εστιάσουμε στη δημιουργία εταιρικών σχέσεων μέσω του εμπορίου με ιδιαίτερη έμφαση στην άμεση γειτονία και στην Αφρική. Επίσης πρέπει να ανοίξουμε τις αγορές, να γίνει πραγματικότητα αυτό για τις επιχειρήσεις οποιοδήποτε μεγέθους. Αυτό σημαίνει ότι οι φυστάμενες συμφωνίες πρέπει να εφαρμοστούν πλήρω και με καλύτερο τρόπο. Τέταρτον, πρέπει να έχουμε τα δυνατότητα, τα μέσα και τα εργαλεία για να μπορεί να είναι δίκαιο και ανοιχτό το εμπόριο και να υπάρχει ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού εντό και εκτό Ένωση. Και πέμπτον, πρέπει να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του εμπορίου, προωθώντα τι αξίε τη Ένωση και εστιάζοντα την κλιματική δράση μαζί με τι προτεραιότητε τη Κομισιόν και τι ανησυχίε του Κοινοβουλίου. Θα αφιερώσω τώρα λίγο χρόνο σε κάθε μια από αυτέ τι πέντε προτεραιότητε το εμπόριο δεν μπορεί να αναδείξει όλο το, το δυναμικό αν δεν υπάρχει σταθερότητα και προβλεψιμότητα. Αυτό μπορεί να υπάρξει μόνο από ένα πολυμερέ σύστημα βασισμένο σε κανόνε. Είπε και η κυρία Φοντρελά, ένα πολυμερέ σύστημα είναι στο DNA τη Ευρώπη. Είναι η αρχή που μα καθοδηγεί στον κόσμο. Η δική μου Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να υποστηρίζει την προσέγγιση ε, και επομένω αυτό σημαίνει ότι η διεθνή τάξη ε, στο πλαίσιο του παγκόσμιου Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου είναι ε, στον πυρήνα αυτό που θα κάνουμε. Σίγουρα υπάρχουν πολλές προκλήσεις. Πρέπει να ε, επικαιροποιηθεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, ε, διότι προσφέρει ένα δρόμο για την επίλυση των εμπορικών ε, ε, αντιπαραθέσεων ε, πρέπει να τον υποστηρίξουμε, αλλά πρέπει και οι κανόνε του να είναι προσαρμοσμένοι στη σημερινή πραγματικότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημαντικό ρόλο και το Κοινοβούλιο για την αντιμετώπιση των δυσκολιών. Αν εκλεγώ, θα κάνω ό,τι μπορώ για να αποτρέψω την κατάρρευση του συστήματος της επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ και να βρω μια συστημική λύση για την μεταρρύθμιση του εφετίου. Επίσης ε, θα συνεργαστώ με τα άλλα μέλη του ΠΟΕ για να αναζωογονηθεί η διαπραγματευτική λειτουργία του οργανισμού. Να εστιάσουμε πρώτα απ' όλα ε, στις ε, διαπραγματεύσεις για τις επιδοτήσεις στην αλληλεία. Είναι ο στόχος 14.6. Επίσης το κανονισμοί για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις εν ώψη της 12ης Υπουργικής Συνέλεσης του ΠΟΕ. Επίσης, θέλω να έχουμε ένα νέο δρόμο για τον ΠΟΕ. Γι' αυτό και θα ετοιμάσω μια πρωτοβουλία για το δεύτερο ήμιση του 20. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε ζητήματα όπως η χρήση των επιδοτήσεων από την Κίνα και άλλους ή την ε, καταναγκαστική μεταφορά τεχνολογίας Επίσης, στα πλαίσια του διεθνού ε, συστήματος ε, υπάρχουν έντονα δείγματα προστατευτισμού από κάποια κράτη. Θα πρέπει εμείς να είμαστε ε, αυτοί που θα μιλήσουμε για ανοιχτό εμπόριο δίκαιο βασισμένο σε κανόνες. Θα είμαι ισχυρός, θα προασπίσω τις, σχέσεις, τις αξίες της Ένωσης εφόσον αυτό χρειαστεί και θα είμαι ένας συνομιλητής που μπορεί να δείξει ηγετική θέση. Η διατλαντική εταιρική σχέση έχει χαράξει ε, και επηρεάσει τις διεθνείς ε, σχέσεις τα τελευταία 70 χρόνια και οι σίγουρα έχουν παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στηρίζοντας αυτό το ανοιχτό σύστημα. Όμως ε, υπάρχουν κάποιες <clears throat> κινήσεις τελευταία που μας ανησυχούν διότι πιστεύουν ότι θα πρέπει βάσει κανόνων να συνεχίσουμε τη σχέση μας. Θα προωθήσουμε τους τομείς κοινού ενδιαφέροντος αλλά πρέπει να μειώσουμε τις εμπορικές εντάσεις όπως ε, είναι στους τομεί που συμφώνησαν ε, ο πρόεδρος Ζήγκερ με τον Τραμπ τον Ιούλιο του 2018. Επίσης ε, θέλουμε να συνεργαστούμε και με άλλες χώρε όπως είναι η Ιαπωνία. Θέλω να είναι θετική η διατλαντική σχέση και να λυθούν το συντομότερο δυνατόν οι διαφορές που έχουμε. Άλλωστε, φέτος το πετύχαμε σε ό,τι αφορά το βόλιο κρέας απαλλαγμένο από ορμόνες και μεταξύ εταίρων αυτά είναι δυνατά. Η σχέση μεταξύ ασφάλειας τεχνολογίας εμπορίου επίσης εξελίσσεται με ταχύς ρυθμούς, επηρεάζει τις σχέσεις μας με όλους τους πρωταγωνιστές. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τις τομείς αυτούς, ιδίως τις ε, τυχέ ασφάλειας ε, των ελέγχων των επενδύσεων και των εξαγωγών. Ε, συμφωνούμε ότι υπάρχουν προκλήσεις λόγω της χρήσης ε, των ε, επιχορηγήσεων από την Κίνα και της, του έντονου κρατικού στοιχείου στην οικονομία της. και θα πρέπει να βρούμε ένα κοινό έδαφο για να συνεργαστούμε με τους ε, εταίρου μας για αυτά τα στρατηγικά ζητήματα. Αλλά και η σχέση μας με την Κίνα είναι ζωτική σημασία, είναι πηγή πλούτου ε, και απασχόλησης. Θα πρέπει όμως να υπάρχει ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού για τις δικές μας επιχειρήσεις, ώστε να μπορούν να ανταγωνιστούν τι κινέζικες και στην Κίνα και στην Ένωση. Αυτό σήμερα δεν συμβαίνει. Θα συνεχίσω τον ε, ενεργό διάλογο. Ε, θα είμαι προσιλωμένο σε τομεί όπω είναι η κλιματική προστασία, περιβαλλοντική προστασία, μεταρρύθμιση του ΠΟΕ και η πειθαρχία σε ό,τι αφορά τι βιομηχανικέ επιδοτήσει. Επίση, θα δώσω προτεραιότητα στι επενδυτικέ διαπραγματεύσει με στόχο την επανεξισορρόπηση των επενδυτικών σχέσεων με την Κίνα. Πρέπει να στηρίξουμε τι αξίε και τα συμφέροντά μα και αντιλαμβάνομαι τι ανησυχίε του Κοινοβουλίου προ αυτό. Η προσέγγιση μα απέναντι στην Κίνα θα πρέπει να επιφέρει μια επανεξισορρόπηση Τη εμπορική σχέση ε, και την αντιμετώπιση των αθέμητων εμπορικών πρακτικών. Θα χρησιμοποιήσω ε, και τα εμπορικά ε, αμυντικά μέσα που έχουμε, γιατί οι σχέσεις μας πρέπει να βασίζονται σε αμοιβαιότητα σε ό,τι αφορά την πρόταση αγορέ, δυνατότητε για του επενδυτέ, για τι επιχειρήσει. Θέλουμε να ενισχύσουμε επίση την ασφάλεια των ε, κρίσιμων υποδομών και τη τεχνολογική βάση, όπω ε, αναφέρει και η ανακοίνωση για την Κίνα του Μαρτίου του 2019. Έχουμε βελτιώσει την εσωτερική εργαλειοθήκη μα ε, με τρόπο είναι ο μηχανισμό για την διαλογή των επενδύσεων, το λεγόμενο screening. Και θα δούμε επίση τι γίνεται με τι ξένε επιδοτήσει στην εσωτερική αγορά και τι στρεβλωτικό αποτέλεσμα μπορεί να έχουν αυτές οι πρακτικές. Θα προωθήσουμε επίσης ε, τις συμφωνίες που έχουμε με τους ε, εταίρους μας ε, από, προς Ανατολάς και με την Τουρκία και με την Ελβετία και με τις χώρες του ΕΟΧ και με την Νότια Μεσόγειο. Βέβαια, σίγουρα πρέπει να αναφέρω και το Brexit εδώ. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα φύγει, προβλέπεται να φύγει από σήμερα στις 31 ημέρες και χωρίς να μπορεί κανείς να προβλέψει ακόμη την τελική έκβαση αν και πολλοί θεωρούν ότι είναι υποχρεωμένοι να προσπαθήσουν να το κάνουν, η Κομισιόν έχει διεξοδικά προετοιμαστεί για ένα Brexit χωρί συμφωνία. Τέλο, η Αφρική πρέπει να είναι προτεραιότητα όλο και περισσότερο. Έχουμε συμφωνήσει πρόσφατα τη Συμμαχία των Συνασπισμών Αφρικής Ευρώπης ε, με βάση ε, μια εταιρική σχέση στις και στις επενδύσεις, ισότιμη σχέση. Αυτό είναι ο δρόμος προς τα εμπρός και έτσι θα συνεχίσουμε. Αφρικανοί ηγέτες και η Ευρωπαϊκή Ένωση από κοινού ε, θα βοηθήσουμε να προωθηθούν οι επενδύσεις. Οι συμφωνίε επίση με Καναδά, Ιαπωνία, Βιετνάμ και πιο πρόσφατα με τη Μερκοσούρ δείχνουν ότι μπορούμε να ασκήσουμε μόχλευση στην εσωτερική αγορά για, την, για το άνοιγμα των αγορών σε παγκόσμιο επίπεδο, να αναδείξουμε του κανόνε τα πρότυπά μα και να βοηθήσουμε να βελτιωθούν κοινωνικέ περιβαλλοντικέ πρακτικέ στι τρίτε χώρε. Θα συνεχίσουμε τι διαπραγματεύσει με Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και θα αναζητήσουμε και νέε εταιρικέ σχέσει εφόσον ε, ευοδοθούν ε, οι συνθήκε. Επίση θα χρειαστεί να εξασφαλίσουμε το πλήρε δυναμικό ε, των συμφωνιών που έχουμε. Θα πρέπει οι εμπορικοί μα εταίροι να σέβονται τι δεσμεύσει του σε όλα τα κεφάλαια Πρέπει επίση να αναβαθμίσουμε τι προσπάθειέ μα για την υλοποίηση ε, και την εφαρμογή των υφιστάμενων συμφωνιών. Έχουμε τον Chief Trade Enforcement Officer. Αυτό θα είναι ένα πολύ σημαντικό ε, σημείο και όποιο αναλάβει αυτή τη θέση θα συνεργαστεί μαζί μου στενά. Θεωρώ επίση πρέπει να κάνουμε και συμφωνώ μαζί σα περισσότερε τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Ε, πάνω από το 80% των ενωσιακών επιχειρήσεων που ασχολούνται με το διεθνέ εμπόριο είναι μικρού και μεσαίου μεγέθου. Υπάρχουν όμω φραγμοί εμπορικοί και επενδυτικοί που του δημιουργούν ιδιαίτερε προκλήσει. Επίση, θέλουμε να τονίσουμε και να προωθήσουμε το δίκαιο ανοιχτό εμπόριο. Πρέπει να αντιταχθούμε στον προστατευτισμό. Πρέπει να προωθήσουμε αμοιβαίε εμπορικέ προποθέσει, δίκαιο ανταγωνισμό με ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού εντό και εκτό, χρησιμοποιώντα εργαλεία παραδείγματο χάρη όπω η Διεθνή Πρωτοβουλία Προμηθειών για αμοιβαιότητα που θα δίνει τη δυνατότητα σε ενωσιακέ επιχειρήσει να επιτύχουν σε διαγωνισμού ε, στο εξωτερικό. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τον αθέμητο ανταγωνισμό αντιμετωπίζοντας πιο αποφασιστικά το πρόβλημα των ξένων επιδοτήσεων που επεράζουν τις ανοσικές επιχειρήσεις και χρησιμοποιώντας και τα μέσα εμπορική άμυνας αλλά και άλλα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Θα ενισχύσουμε βέβαια και την εργαλειοθήκη μας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε παράνομα και διακριτικά εμπορικά μέτρα από τρίτες χώρες όταν δεν μπορούμε να προσφύγουμε στον ΠΟΕ. Πρέπει να είναι όμως το εμπόριο και βιώσιμο, όχι μόνο δίκαιο και ανοιχτό. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε παγκόσμιες προκλήσεις όπως κλιματική αλλαγή. Πρέπει να προστατεύσουμε το περιβάλλον, να ενισχύσουμε τα εργασιακά πρότυπα. Γι' αυτό τα κεφάλαια βιώσιμη ανάπτυξη, όλε τι συμφωνίε ε, είναι πάρα πολύ σημαντικά, καθότι περιλαμβάνουν και δεσμευτικέ ε, ε, διατάξει για το περιβάλλον και την εργασία. Θα κάνω χρήση για την επίτευξη αυτών των στόχων όλων των δυνατοτήτων που μου δίνει η εργαλειοφυκή που έχουμε στη διάθεσή μα. Εμπορικέ προτιμήσει, διμερεί εμπορικέ συμφωνίε, πολυμερεί δράσει. Αν εκλεγώ, θα συνεργαστώ μαζί σα και για να βελτιώσουμε το γενικευμένο σύστημα προτιμήσεων να ε, το ανανεώσουμε. Είναι αυτό που δίνει προτιμησιακή ε, πρόσβαση στις εξαγωγές ε, για αναπτυσσόμενες και λιγότερα ανεπτυγμένες χώρες. Οι εταίροι μας θα πρέπει να μπορούν να έχουν τα κίνητρα για να προχωρήσουν προς τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω αναπτυξιακών πολιτικών εστιάζουμε περισσότερο στο κλίμα και τη βιωσιμότητα, γιατί ακριβώ αυτό θέλουν οι πολίτε. Και οι αξίε αυτέ θα ενσωματωθούν στο εμπορικό θεματολόγιο. Αξιότιμοι ότι με βουλευτέ, η εμπορική πολιτική είναι από τι πιο δυναμικέ ε, πολιτικέ. Έχουμε σημαντικό θεματολόγιο. Είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για το πολυμέρε σύστημα. Έχουμε ένα εύθραυστο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα. Το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή σα από την Συνδίκη τη Λισαβόνα έχουν αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο για τη χάραξη του εμπορικού θεματολογίου. Θα συνεργαστώ μαζί σα η Ευρώπη πρέπει να είναι ο παγκόσμιο πρωταθλητή ενό δίκαιου βιώσιμου εμπορίου που βασίζεται σε κανόνε. Ελπίζω με τη βοήθειά σα να ενισχύσουμε αυτό τον ηγετικό μα ρόλο. Μπορούμε να δράσουμε και να δώσουμε αποτελέσματα. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χόγκεν, λέει ο πρόεδρο. Και τώρα ακολουθεί ο πρώτο γύρο ερωτήσεων από του συντονιστέ των πολιτικών ομάδων. Και ο πρώτο πρόκειται από το έλκυνε ο Κριστόφ Χάνσεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε Επίτροπε και κύριε υποψήφιοι Επίτροπε. Εμείς και οι έχουν πιο μεγάλη μορική Ολοκλήρωση, Μιλούμε για 6 εκατομμύρια θέσει απασχόληση, το 1 τρίτον του παγκοσμίου ΑΕΠ, το οποίο δημιουργείται όμω αυτή τη στιγμή η πολιτική που ακολουθεί η Αμερικανική κυβέρνηση με αυτού του μονομερεί κινήσει με του δασμού έχει ταράξει το, τον ΠΟΕ που είναι ο πυλώνα του Διεθνού Εμπορίου. Οπότε σα ρωτώ, εσεί πρόκειται να φέρετε κάποιε διορθωτικέ κινήσει στη σχέση με τι ΗΠΑ ε, και πρόκειται να υποστηρίξετε το παγκόσμιο ε, εμπόριο ε, και όλα αυτά κόντρα στον Πρόεδρο, ο οποίο έχει φέρει αυτή την υπονόμευση τόσο καιρό τη παγκόσμια σταθερότητα σε αυτό το επίπεδο. Κύριε Χόγκεν, έχετε το λόγο. τις στιγμές της μεγάλης έντασης. Δεν θα πρέπει να χάνουμε αυτού του, την συνολική εικόνα, γιατί έχουμε 3 εκατομμύρια συναλλαγέ σήμερα με τη είπα και η σχέση μας με τη χώρα αυτή είναι πιο μεγάλη, πιο βαθιά, πιο σημαντική εμπορική σχέση. Και υπάρχουν οι βάσεις επομένως να πάμε καλύτερα. Είχε γίνει συνάντηση τον Ιούλιο του 2018 μεταξύ Γιούνκερ και του Πρόεδρου των ΗΠΑ, αλλά δεν ε, υπήρξε μεγάλη πρόταση από τότε. Οπότε η νέα πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή Φοντερ Λάγεν έχει έναν στόχο που για τον πρέπει να σας πω ότι να αρχίσει ένα θετικό θεματολόγιο και ότι θα πρέπει να κινηθούμε με τη ΣΥΠΑ προς ε, ε, κάποια αμοιβαία υποφιλή σχέση. Αλλά βέβαια χρειάζονται δύο για μια συνεργασία και δύο πλευρές. Οπότε θα πρέπει να δούμε γιατί ε, έχουν αργήσει τόσο πολλοί Αμερικανοί να κάνουν μια κίνηση, αλλά θα πρέπει αυτό να γίνει με έναν τιμιο τρόπο και Επομένως, ε, το σημαντικό είναι τώρα να δούμε τη διάσταση των πραγμάτων που φέρει για τους δύο και έγινε πρόσφατα ε, η συμφωνία για το βόλιο κρέας τον Ιούλιο και πρόκειται για ένα ξεκάθαρο σημείο που δείχνει ότι εμείς προτιθέμεθα να υπάρχει διάλογος και συνεργασία. Η δε σχέση μεταξύ ασφάλειας, τεχνολογίας και εμπορίου είναι μια σχέση που εξελίσσεται συνεχώς, οπότε χρειαζόμαστε τις ε, είπα ε, για τον ΠΟΕ, ούτως ώστε στον ΠΟΕ να εξασφαλίσουμε όλα αυτά και θα πρέπει να επισημάνουμε αυτά τα θέματα που τους ενδιαφέρουν. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται Επίσης ε, για όλες αυτές τις ε, κρατικές επιδοτήσεις που ξέρουμε ποια χώρα τις κάνει και θα πρέπει επομένως ε, ε, όλο αυτό το θεματολόγιο να προωθηθεί σε μια κατάσταση κλειστής αγοράς και άρα θα πρέπει να συνεργαστούμε για όλα αυτά. Αλλά όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν υπό την αιγίδα του ΠΟΕ. Οπότε όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν με γνώμονα το κοινό συμφέρον. Άρα θα πρέπει να οδηγηθούμε σε συμφωνίες που ωφελούν και τις δύο πλευρές. Έτσι βλέπω τα θέματα. Παρακάτω. Ναι, ναι, έχω και μια επερώτηση. Αυτή τη στιγμή, ξέρετε, σήμερα ή αύριο, ο ΠΟΕ πρόκειται να κρίνει για μια υπόθεση που έχει υποβληθεί και έχουμε δει ήδη τα θέματα στα οποία θα πιέσουν οι ε, ΙΠΑ, ε, ελιές, κρασί και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει όσον αφορά την ε, προμήθεια των Οπότε, μήπως έτσι θα διασπαστεί η ενιαία στάση των κρατών μελών. Γιατί αφού έχουμε στο επίκεντρο γεωργικά προϊόντα, πώς αυτό θα επηρεάσει τον τομέα της γεωργίας. Η Επίτροπος, μάλλον τον λέει ο υποψηφίος Επίτροπος, έχει προτείνει μια ε, λύση σε σχέση με την υπόθεση αυτήν, δηλαδή να συμμορφωθεί πλήρως η έργος. Αλλά υπάρχει και άλλη υπόθεση που εκκρεμεί στον ΠΟΕ, που αφορά τις ΠΟΕ. Είναι η Boeing. Και κάποια στιγμή θα κρατήσει αυτή Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προτείνει κάποιες θετικές λύσεις για αυτό το πρόβλημα που έχουμε να λύσουμε. Έχουμε τα αντίπεινα, τον είπα, τα οποία ενδεχομένω ακολουθήσουν οι άνοιοι είναι δεσμένες. Οπότε εμείς προσπαθούμε να βρούμε πεδίο συνεννόησης, αλλά ακόμα αυτό δεν το έχουμε πετύχει. Και είναι κατανοητή η δυσκολία για όλα αυτά τα προϊόντα που κρίνονται αλλά ας περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασιστεί, τι θα κάνουν οι όσον αφορά τα αντίπεινα. Πάντως εμείς θα πρέπει να προωθήσουμε τα συμφέροντά μας και θα πρέπει επίσης να προωθήσουμε τα δικά μας συμφέροντα. Για τους Σοσιαλιστές Δημοκράτες, η κυρία Καθλίν Φαν Μπρέμπτ. This Σαμποτάζε πάθε το μικροφώνο μου, λέει η κυρία Φανμπρέμπτ. Δουλεύει. another one. Χρησιμοποιήστε άλλο μικρόφωνο, προτείνει ο πρόεδρος. Now even further away, Commissioner, but that's... Απομακρυνθήκαμε λίγο, αλλά μόνο, μόνο σε απόσταση. Δεν έχει συμβολική σημασία. Κύριε υποψήφιε ε, επίτροπε και κύριε επίτροπε, έχω δύο συγκεκριμένε ερωτήσει όσον αφορά τι ε, συμφωνίε ελευθέρου εμπορίου. Πρώτα, πρώτα. Για τα πρότυπα TST. Τι έγινε με την Νότια Κορέα, τι έγινε με την Κολομβία, είδατε ότι πέρσι είχαμε 169 νεκρούς από ακτιβιστές περί ανθρωπινών δικαιωμάτων πέρσι. Άρα δεν πάνε καλά τα πράγματα. Θα πρέπει είπαμε, ε, να χρησιμοποιήσουμε ό,τι μπορούμε όσον αφορά τον στόχο μα για το κλίμα κλπ. Το θέμα είναι πώ θα γίνει αυτό στην πράξη. Αν δεν κάνει το ε, πώς το DST σήμερα. Η Επιτροπή είχε συγκεκριμένα 15 πώ ήταν προγράμματα δράσης, ε, κάποια από αυτά δεν θεωρείτε ότι δεν αποδίδουν και θα πρέπει κάτι να κάνετε, να τα βελτιώσετε, να βρείτε καινούργια εργαλεία, καινούργια μέσα. Τι γίνεται επίσης, διακόπτει. Διακόπτει ο πρώτος και λέει αυτά στην επερώτησή σας που μπορείτε να κάνετε, ο Επίτροπος. Ευχαριστώ κύριε Φανμπρέμ Ξέρω το θέμα. από τους συναδέλφους σας, από τους συντονιστές σας που θέλετε να έχουμε καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά την υλοποίηση των ισχυωσών συμφωνιών. Και το παράδειγμα με την Κόρεα μας οδηγεί στο ότι για πρώτη φορά χρησιμοποιούνται αυτοί οι μηχανισμοί επίλυσης διαφορών ούτως ώστε να συμμορφωθεί η χώρα αυτή με όσα δεν τηρούσε. Άρα να, μια δοκιμή. Για πρώτη φορά δούμε τι γίνεται όσον αφορά εφαρμογή υλοποίηση με κάποιον ε, εταίρο μας. Να δούμε εάν θα κάνουν αυτά που έκαναν όταν προσυπερέψαν τη συμφωνία. Και πρέπει αυτό να το μεταλλευτούμε και έχουμε αυτό το πρόγραμμα δράσης. Έχουμε και το θέμα της επίλυσης διαφόρων. Είναι σημαντικό για την κοινωνία των πολιτών, σημαντικό για τις ε, θεσμικές ρυθμίσεις εδώ της Ένωσης Άρα θα πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω ευκαιρίε ούτω ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε, να υποστηρίξουμε και οικονομικά τις καταγγελίες, να βρεθούν τα αποδεικτικά στοιχεία ούτω ώστε να ε, πλαισιωθεί, να είναι βάσιμη μια υπόθεση. Άρα περιμένουμε να γίνει η πλήρης εφαρμογή και αυτό θα το δούμε. Αυτό το τεστ, αυτή τη δοκιμή που αποτελεί η Κορέα. Φανμπραντεύ ερώτησε, ναι, σε σχέση με την απάντησή σα Για κοιτάξτε, τι γίνεται στην Βραζιλία. Τι έγινε το καλοκαίρι φέτο, τα συζητήσαμε ήδη. Τι γίνεται με τη Συμφωνία Μερικοσούρ. Πολλοί λένε ότι η συμφωνία αυτή, εάν σήμερα ίσχυε, τότε θα είχε σωθεί ο Αμαζόνιο. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι χρειάζονται αυτέ οι συνδικές οι προ... προκύρωσης τέλος πάντων. Και αυτό θα έπρεπε να γίνει και στο Μερικοσούρ πριν αρχίσει η διαδικασία της ακύρωση Εσείς σύμφωνα με αυτή την άποψη γιατί εν τη αυτή η περιπτώση θα είχαμε ακόμα ένα όπλο για να εξασφαλίσουμε ότι θα κατοχυρωθούν όλα αυτά που είπατε στην εισήγησή σας. Θα εξασφαλίζαμε ότι θα υπήρχε πραγματική δέσμευση προς την κατεύθυνση τη Συμφωνία των Παρισιών. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, επομένω για τη φάση πριν την κύρωση. Κύριος ο πρόεδρος Μπολσονάρο αλλιώ τα έλεγε πριν εκλεγεί πρόεδρος. Και πάντα στην πολιτική έτσι γίνονται. Αφού εξελέγει λοιπόν, αποφάσισε να αλλάξει στρατηγική. Και σήμερα με συμφωνία των Παρισίων μιλούμε για 12 εκατομμύρια εκτάρια που θα έχουν αναδάσωση Με το 2030. Είπαμε για δέσμευση καλύτερη διαχείριση των δασών. Αν δεν υπήρχε η εμπορική πολιτική και η συμφωνία, πώς θα πιέζαμε τις χώρες της συμφωνίας Μέρκοσουρ και την Βραζιλία. Όλοι φρικιάσαμε αυτό που έγινε στον Αμαζόνιο, αλλά δεν μπορούμε τώρα να κάνουμε τίποτα. Δεν έχουμε τα μέσα χωρίς να βοηθήσει η εμπορική πολιτική. Οπότε στην ε, τελική ευθεία της κύρωσης τότε είμαστε πιο δυνατοί. Ξέρω τι εννοείται με τη φάση πριν την κύρωση, αλλά προσοχή. Γιατί σε μια τέτοια προβληματική θα ζητήσουν, μια που μιλούμε για εμπόριο, να ανοίξουμε κι εμείς και άλλα κεφάλαια. Και τώρα η Κάριν Κάρλς Μπρο. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ για την ε, εισήγησή σα. Θα πρέπει να υπάρχει ισότητα ανταγωνισμού για όλε τι εταιρείε, σε όλε τι χώρε, τόσο ώστε να μπορούν να ανταγωνιστούν στο παγκόσμια σκηνή. Αυτό θα πρέπει να είναι βασικό για το ψηφιακή εμπόριο. Εσεί τι θα κάνετε ούτως ώστε να βοηθήσετε να υπάρχει μια τέτοια ισότιμη ε, ψηφιακή οικονομία για αμοιβαιότητα, ισότητα ανταγωνισμού, ε, προς του καταναλωτή και όλοι να ωφελούνται και οι επιχειρήσεις αλλά και ο κόσμος εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα πώς θα εξασφαλίσετε ότι όλα αυτά τα οποία προβλέπονται μέχρι τώρα για το ηλεκτρονικό εμπόριο θα βοηθήσουν τόσο ώστε να έχουμε ένα πλαίσιο συνεπές δίκαιο για το διεθνέ εμπόριο. Και όταν παρουσιάσατε τη στρατηγική σας ως Επιτροπή, πότε θα το ολοκληρώσετε Ο κύριο ε, Ναι, ναι, ευχαριστώ. Βεβαίω θα πρέπει να είναι δίκαιο, ανοιχτό το εμπόριο, να υπάρχουν παγκοσμίοι κανόνε. Αυτό και ακριβώ λέμε για τι ΗΠΑ. Και ο Ρομπέρτα Ζεβέδο από τον ΠΟΕ σήμερα ήρθε και τα συζητήσαμε να δούμε τι θα κάνουμε και θα ήθελα να δείξουμε πιο ηγετική στάση στο μέλλον και θα συνεργαστούμε στενά μαζί του για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να έχουμε τέτοιους κανόνες για το διεθνές εμπόριο ε, πολυμερές και δίκαιο και ανοιχτό στα πλαίσια του ΠΟΕ και όπως τα έχουμε συζητήσει εδώ πολλές φορές να δούμε πώς θα προστατεύσουμε εαυτούς μέσω του εμπορίου. Επομένως, για τις ε, επιχειρήσεις ε, προκινούμεθα πολύ προσεκτικά, το ίδιο και για τις κρατικές συμβάσεις και το Συμβούλιο επίσης στο ίδιο μήκος κύματος, μίλησα με τον Υπουργό Οικονομίας της Γερμανίας πρόσφατα και επίσης ε, ψάχνουμε ακόμα να δούμε πώς θα προσεγγίσουμε τις γερμανικές θέσεις. Πάρα πολύ σημαντικό ότι θα γίνει στην αγορά, την ηλεκτρονική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχουμε επομένω κάποιο μέσο, ούτως ώστε να δούμε τι θα κάνουμε όσον αφορά τις επιδοτήσεις κάτι το οποίο το μετέρχεται η Κίνα για να ωφεληθεί από τη δική μας αγορά. Εμείς είμαστε περήφανοι γιατί έχουμε εσωτερική αγορά ανοιχτή, με οικονομία της αγοράς, αλλά πάρα πολλές φορές κάποιοι καταχρώνται, εκμεταλλεύονται αυτό μας το χαρακτηριστικό. Επομένως θα πρέπει να έχουμε γερή άμυνα όταν χρειάζεται. από 140 προσφυγέ των εταιρείε σχετίζονται με μια συγκεκριμένη χώρα και επομένως χρειαζόμαστε να υπάρχουν τα μέσα και να ισχύουν για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα φαινόμενα γιατί αλλιώς δεν ωφελούν δεν πρόκειται να μας οδηγήσουν στον επιθυμητό στόχο άρα κάποιες τεχνολογίες κάποια δέστετα προϊόντα μα όντω πρέπει να προστατευτούν και αυτό είναι όλο ένα και πιο σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ για την απάντησή σας. Τώρα ε, στην επερώτηση λέει. Κύριε, όσον αφορά τα ψηφιακά, είδαμε ακριβώ ότι έχουν δημιουργήσει προστριβέ και οπότε να δούμε πώ θα έχουμε σωστό προβληματισμό, ε, μην έχουμε προστριβέ. Άρα, εσεί τι θα κάνετε, πώ θα εμπλακεί η, η κοινωνία, για να έχουμε σωστή αξιολόγηση, υποπτία, πώς θα βελτιώσετε την επικοινωνία για τις εμπορικές συμφωνίες. Και έτσι όλοι να καταλάβουν πόσο ωφελεί το εμπόριο. Ναι, με χαρά μου να εμπλακούν όλοι, όλοι αυτοί οι παράγοντες. Εθνικά Κοινοβούλια, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Κοινωνία. Ναι, αυτό είναι προτεραιότητα για να έχουμε μια ενιαία ψηφιακή αγορά και την προσπάθεια ετών αυτή. Αλλά πάμε σιγά σιγά. Χρειάζεται ένα τοπίο ισοτιμίας. Και μέσω του ΠΟΕ προσπαθούμε ότι θα γίνει και με την Κίνα. Για να ολοκληρωθούν οι συνομιλίες για το ηλεκτρονικό εμπόριο, με τι θα γίνει με τη στρατηγική, με αυτό το θεματολόγιο για τα ψηφιακά, όχι μόνο σε επίπεδο Ευρώπη, αλλά παγκόσμια και να ισχύσει το πλαίσιο που επιβάλλεται. Άρα, έτσι πρέπει να προβάλλουμε τις ευεργετικές συνέπειες του εμπορίου. Δεν είναι πάντα εύκολο να κάνουμε ό,τι μπορούμε το ώστε να υπάρχει σωστή ενημέρωση. Σε αυτό να βοηθήσουμε. Και τώρα, Χάιντι Χάουτολα για ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Υποψήφιοι Επίτροπε, καλησπέρα. Είδα κάτι εκεί στις γραπτές απαντήσεις. Ε, λέτε ότι θα έχετε μηδενική ανοχή στην παιδική εργασία. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να κοιτάξετε διάφορα ψηφίσματα της Επιτροπής μας όπου ζητάμε την υποχρεωτική δέουσα επιμέλεια στην περίπτωση παραβίασης ε, των θεμελιωδών δικαιωμάτων από ευρωπαϊκές εταιρείες ή στην περίπτωση αποδάσωσης. Και ευχαριστώ να σας πω πως ε, η Κομισιόν ε, τον Ιούλιο αποφάσισε για ρυθμιστικά και μη ρυθμιστικά μέτρα για να καταπολεμήσουμε την αποδάσωση στην αλυσίδα προμηθειών. Ποια θα ήταν η δική σας η προσέγγιση αν ε, ε, κληθείτε να συμμετάσχετε σε προσπάθεια να ε, τεθεί το θέμα αυτό της υποχρεωτικής δέουσας επιμήλειας στην εφοδιαστική αλυσίδα. Σας ευχαριστώ κύριε Χάτουλα. Αντιλαμβάνομαι ότι η Επιτροπή αυτή έχει το δικαίωμα της νομοθετικής πρωτοβουλίας, κατά το οποίο ανέφερε και η κυρία Φαντερ Λάιν και το οποίο και εγώ στηρίζω. Οπότε αναμένω τη συνεργασία με την Επιτροπή σας, αν αυτό γίνει η προτεραιότητα της Επιτροπής σας για οποιαδήποτε τεχνική στήριξη, ακροάσεις, εκθέσεις ή οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί. Οι υπηρεσίε μου θα είναι στην διάθεσή σας και ελπίζω να σας βοηθήσουν. Επίσης έχουμε και ένα καλό ιστορικό όσον αφορά τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παραδείγματο χάρη ο κανονισμός περί ορυκτών από περιοχές ε, με σύγκρουση. Έχουμε και τον κανονισμό περί ξυλίας ε, που επίσης ε, απαγορεύει την εμπορία ξυλίας από τέτοιες περιοχές. Έχουμε επίσης την οδηγία για επανόρθωση στα θύματα και το άλλο θέμα βέβαια αφορά την οδηγία αφορά τις ε, εκθέσεις για τις ε, έξι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές ε, εταιρείες και οπωσδήποτε μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Αλλά οπωσδήποτε θεωρώ ότι είναι μια καλή αφετηρία. Και βεβαίω η εμπορική πολιτική μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλα ζητήματα την ισότητα των φίλων. Αν αποφασίσετε λοιπόν να ξεκινήσετε με νομοθετική πρωτοβουλία. Εγώ ευχαρίστω θα την υποστηρίξω. Σας ευχαριστώ. Έχετε και επερώτηση. Σας ευχαριστώ. Ανακάλυψα επίσης τι γραπτές απαντήσεις σα πολλές αναφορές στην εφαρμογή των στόχων της ε, βιώσιμη ανάπτυξη. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω πώς θεωρείτε ότι η Κομισιόν θα πρέπει να καθορίσει τις ε, προτεραιότητες της. Ε, θεωρείτε ότι θα πρέπει να τα κάνει αυτά η ίδια η πρόεδρος ή πώς αλλιώς. Και εσείς συγκεκριμένα παρακαλώ πώς θα συνεισφέρετε. Νομίζω πως τώρα είναι ευκαιρία να μιλήσουμε για τον επικεφαλής ε, συμμόρφωσης που έχουμε κατά νου. Και τα έχει πει η κυρία Φεντερλάιν ότι είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Θα ήθελα λοιπόν να το προχωρήσουμε αυτό το στομότερο δυνατόν το 2020 πρέπει η Επιτροπή και εγώ να είμαστε σε επαφή με όλους τους ενδιαφερόμενους, να δούμε ποια είναι τα κριτήρια αναφοράς ε, που θα μπορέσουμε να έχουμε για την ε, αυτή θέση που θα πρέπει βεβαίως να είναι πολιτικά υπόλογος αλλά και σε αρκετά υψηλό επίπεδο για να έχουμε αρκετά καλή επικοινωνία και ένα καλό επίπεδο εφαρμογής ε, και επιβολής. Όπως είπα και στην κυρία Φαν πιο πριν, η εμπορική πολιτική και οι βιώσιμοι στόχοι θα πρέπει να πηγαίνουν χέρι με χέρι. Πρέπει λοιπόν να τα στηρίξουμε πλήρω. Θεωρώ ότι πρόκειται για μια καλή πρωτοβουλία και αναμένω να την συζητήσουμε. Σα ευχαριστώ. Τώρα για το IDO Macros Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υποψήφιε Επίτροπε. είναι νομίζω αντικείμενο συνένεσης ε, πως δεν θέλουμε κάποιο εμπόριο λεσέφερ. Χιλιάδες ε, πολίτες είχαν κατά τους δρόμους κατά τη ΣΕΤΑ και της ε, συνθήκης TTIP. Ένα βασικό θέμα τότε ήταν η κατάσταση των αγροτών μας, αλλά και άλλων κατηγοριών. Εν της ασφάλειας ε, των καταναλωτών και της διατροφικής ασφάλειας. Ε, τώρα έχουμε μπροστά μας την Μερκοσούρ. Δεν ξέρουμε όμως ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Με βάση ποια μελέτη αντικτύπου εργάστηκε η Κομισιόν. Γιατί υπάρχει υποψία ότι την στιγμή της ε, σύναψης της συμφωνίας τον Ιούνιο δεν ήταν σαφείς οι πιθανές επιπτώσεις για τους αγρότες μας. Κύριε Χόγκαν, τι θα κάνετε με τη συμφωνία του Μερκοσούρ εάν η νέα μελέτη αντικτύπων δείξει μεγαλύτερους δυνητικούς αντικτύπους στην Γεωργία από ό,τι φοβόμαστε μέχρι στιγμής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντιλαμβάνομαι βέβαιως τις ανησυχίες που υπάρχουν για την συμφωνία με το Μερκοσούρ. Ε, βεβαίως, πρέπει να γίνουν κάποιες ε, παραχωρήσεις Κανείς, ε, γεωργός δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένο. Αλλά αν δείτε σωρευτικά το τι έχουμε επιτύχει ε, με τις εμπορικές συμφωνίες, θα δείτε ότι είναι πολύ θετικό το αποτέλεσμα ε, γενικά για τη Γεωργία. Σε σχέση με τη ΣΥΤΑ, σε σχέση με την Ιαπωνία, το Μεξικό, έχουμε πολύ θετικά αποτελέσματα. Η συμφωνία με τη Μερκοσούρ είναι οπωσδήποτε μια συμφωνία για την οποία θα γίνει μια μελέτη αντικτύπου βιωσιμότητας ε, και θα κάνουμε και μια σορευτική μελέτη αντικτύπου για το τι σημαίνουν όλες αυτές οι συμφωνίες για τους ε, γεωργούς. Οπότε, με το να κρατάμε τις ποσοστό στο δυνατόν πιο χαμηλές ε, για το βόλιο κρέας, τη ζάχαρη, την εθανολή, τα πουλερικά, νομίζω ότι έχουμε επιτύχει ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα, το οποίο βεβαίως αφορά όλους τους ε, κλάδους σε σχέση με το ότι έχουμε επιτύχει στο Mercosur. Η ανάλυση λοιπόν που ζητάτε για το τι μπορούμε να σας δώσουμε για το 2020-2021 πριν φτάσουμε στην κύρωση αυτής της ε, συμφωνίας για να μπορέσουμε να έχουμε κάποια θετικά αποτελέσματα, όπως παραδείγματο χάρη στην τομέα των γαλακτοκομικών από βουτυρωμένο γάλακτο σε σκόνη και ε, το κρασίου και άλλο, όπου θα πρέπει να επιμείνουμε σε μια ποσόστοση με σημαντικές δικλίδες ε, ασφαλείας, ε, όπου θα έχουμε ένα μηχανισμό διασφάλισης για πρώτη φορά σε σχέση με μια ποσόστοση δασμών. Δηλαδή, αν υπάρξει απότομη αύξηση των εισαγωγών με βάση τα στοιχεία, μπορούμε να αποσύρουμε την ε, συγκεκριμένη αυτή ποσόστο για μια περίοδο μέχρι 4 έτη. Είναι αυτά δικλείδε ασφαλεία που για πρώτη φορά υπάρχουν. Κύριε Μπουφαλτά, ναι. έχετε και άλλη ερώτηση. Ευχαριστώ. Μετά, τον Ιούνιο υποσχεθήκατε ένα δισεκατομμύριο ευρώ στους αγρότες μας ως βοήθεια. Από πού προέκυψε αυτός ο αριθμός, τι ήτανε, είπατε κάτι για, να πείτε για δημόσιες σχέσεις ή ε, ελπίζετε ότι θα μείνει. Ε, ε, Εκπλήσω με που αμφισβητείτε τις επιδοτήσεις προς τους αγρότες. Ε, δεν έχω ακούσει κανένα αγρότη να είναι εναντίον, αλλά πρόκειται για κονδύλια τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στην περίπτωση ανισορροπίας της αγοράς και ήταν κάτι το οποίο είχε συζητηθεί τότε με τον πρόεδρο της Κομισιόν για να διασφαλίσουμε τους κλάδους μας που ασχολούνται σε κάποιο με κάποια ζητήματα όπου ήμασταν θα έλεγα στην άμυνα ότι θα υπάρχουν ήδη κλείς για την ποιότητα των ε, προϊόντων και είναι εκτός του προπολογισμού της ΚΑΠ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνάμε τώρα στο ECR Get Bourgeois. Ευχαριστώ. εμεί υποστηρίζουμε βέβαια το δίκαιο εμπόριο ως βασί διαλόγου αλλά και ανάπτυξης. Γι' αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε σύγχρονες εμπορικές συμφωνίες, να υπερασπιστούμε την πολυμερή προσέγγιση και τον ΠΟΕ, αλλά να βεβαίως να προστατεύσουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση από τον ντάμπινγκ αφενός αφετέρου, όποτε κατηγορούμαστε αδίκωση για dumping στο εξωτερικό, όπως συμβαίνει παραδείγματος χάρη με τις ε, πατάτες, ε, πρώτα στη Νότια Αφρική, τώρα κάποιες χώρες της Νότιου Αμερικής. Ε, θα πρέπει λοιπόν να δράσουμε γιατί δεν δρούμε αρκετά γρήγορα και αποφασιστικά. Είστε έτοιμος να προστατεύσετε τις επιχειρήσεις μας, τις θέσεις εργασίας. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με τα όσα είπατε. Πρέπει να είμαστε πράγματι ταχύτεροι και πρέπει να είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βέβαια, πρέπει να έχουμε τις απαραίτητες ενδείξεις, αποδείξει ότι μπορούμε πράγματι να δράσουμε έτσι και να τους βοηθήσουμε σε περίπτωση που υπάρχουν κάποιοι ισχυρισμοί σε βάρος τους, γιατί το ξέρετε φαντάζομαι και εσείς ε, από τη Φλάνδρα Υπάρχουν ε, μικρές επιχειρήσεις που δεν μπορούν οικονομικά να επεξέλθουν στο κόστος μιας χρονοβόρας δικαστικής διαμάχης. Επομένως, αυτό το οποίο εμείς ε, εντατικά στη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Trade ε, αναζητούμε είναι να μπορεί να γίνεται νωρίτερα η επίλυση και επίσης ε, τώρα μπορούμε να κάνουμε περισσότερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τους παρέχουμε υποστήριξη, βοήθεια και σε συγκεκριμένε περιφέρειες και κράτη-μέλη. Δεν θέλουμε να υπάρχει αλληλεπικάλυψη και εστιάζουμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αν δεν έχουν την απαιτούμενη υποστήριξη σε εθνικό επίπεδο. Ε, δεν ξέρω αν γνωρίζετε τι επέβαλε η Κολομβία, δηλαδή κάποιους δασμούς, ε, ιδίως ε, στις βελγικές πατάτες. Νομίζω γι' αυτό μιλήσατε. Εγώ μίλησα με τον Υπουργό των Αρμόδιων της Κολομβίας, συγκεκριμένα τον συνάντησα πέρυσι, αλλά δεν έχουμε ακόμη καταφέρει ε, να επιλύσουμε με ένα θετικό τρόπο αυτό το ζήτημα, άρα θα πρέπει να στήσουμε άλλες επιλογές. Πρόεδρος, έχετε δεύτερη ερώτηση. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι πρέπει να κινηθούμε γρήγορα. Γιατί βλέπετε τώρα εξαπλώνεται το φαινόμενο. Πρώτα η ότι Αφρική, τώρα είναι οι Αμερικανικές χώρες. Συγκεκριμένα λοιπόν θεωρείτε ότι ο Chief Trading Informant Officer θα μπορεί να παρεμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Νομίζω ότι θα έχει πολλή δουλειά να κάνει. Αυτό είναι σαφές. Και είναι καλό αυτό βέβαια. Αλλιώ θα πρέπει να τα κάνει όλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά θα εργαστούμε μαζί για να υπάρξει σωστό επιμερισμό εργασία και να έχουμε την καλύτερη δυνατή έκβαση. Κύριε Μπουρζουά, για να σα καθησυχάσω, το ζήτημα που γνωρίζω ότι σα απασχολεί για τι βελικέ πατάτε ε, και σίγουρα είναι ένα προϊόν που χαρακτηρίζει, είναι το σύμβολο τη χώρα, είναι ένα θέμα που μα απασχολεί πάρα πολύ σοβαρά. Φαντάζομαι και την κυρία Φαμπρέμ την ενδιαφέρει πολύ. Και πρέπει να σας πω ότι έχουμε υποβάλει ένα αίτημα για αναθεώρηση ε, της απόφασης ε, των Κολομβιανών αρχών. Δεν καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εξιολογούμε τώρα την κατάσταση. Υπάρχει και αυτό, αυτή η ε, διασκαστική διαμάχη σε επίπεδο ΠΟΕ με την Κολομβία. Και οι γερμανικές πατάτες. Δεν είναι μόνο οι βελγικές πατάτες, λέει ο πρόεδρος, και τελευταίος συντονιστής από την ΚΟΕ, ο Χέλμουντ Σόλτς. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα κύριε Χόγκαν. Εδώ είμαι κύριε Επίτροπε. Μιλάμε για κανόνες, για δίκαιο ανοιχτό εμπόριο, για τις αρχές, για την εφαρμογή και στη γραπτές σας απαντήσεις Είπατε ότι θα προσπαθήσετε να βρεθεί μια λύση και στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Θέλετε μια νέα ισορροπία εκεί με τη δημιουργία εφόσον χρειάζεται νέων κανόνων για ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού. Και αναφέρεται κάπου και το πολυμερές σύστημα. Έχουμε την ε, αρχή της Γενέβης ε, και έχουμε την Παγκόσμια Πράσινη Συμφωνία. Και το ένα είναι ότι θα πρέπει ο στόχος να είναι η οικονομική και κοινωνική σταθερότητα, η ευημερία, η περιβαλλοντική αηφορία και βιωσιμότητα. και μια ισορροπία να μην υπάρχει δηλαδή πρωτοκαθεδρία των πιο ισχυρών. Αυτή η αρχή ε, τη δέουσα επιμέλεια, παραδείγματο χάρη, για την αλυσίδα εφοδιασμού που προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι ένα εργαλείο που θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε. Σε μια απάντηση που έδωσα πιο πριν, λέει ο κύριο Χόγκαν, είπα πω αν το αποφασίσει η Επιτροπή σα ε, και δώσει προτεραιότητα σε αυτή την πρωτοβουλία για τη δέωση επιμέλεια στο πλαίσιο του προγράμματο εργασία και στο πλαίσιο ανάληψης πρωτοβουλίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, και αν αυτή η γραμμή ε, υιοθετηθεί και από την κυρία Φοντρελάν, με τα χαρά θα ακολουθήσω τι ε, τις προτάσεις σας, λαμβάνοντας υπόψη και την εμπειρία που έχουμε σε ορισμένου από αυτού του τομεί. όπω είναι τα υφάσματα και τα Είδαμε τι έγινε με ΙΠΑ και Γουατεμάλα, για παράδειγμα. Χρειάστηκαν 7 χρόνια και η υπόθεση δεν έλξε με τον ιδανικότερο τρόπο. Είμαι ανοιχτό σε υποδείξεις ε, και σίγουρα θα ακούσω τις δικές σας απόψεις και θα δούμε πώς μπορούμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή έκβαση. Σίγουρα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ενίοτε δεν λειτουργεί όπως θέλαμε και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, να μελετήσουμε όλες αυτές τις υποθέσεις. Υπάρχει δεύτερη ερώτηση. Ναι, πώς θα γίνουν όλα αυτά δεσμευτικά και πώς θα εφαρμόζονται στην πράξη. Για παράδειγμα, χρειάζεται υποστήριξη και από τους διαφερομένους ε, φορείς και από τους καταναλωτές, γιατί το εμπόριο σημαίνει τρόπος παραγωγής κατανάλωση, ένας τρόπος ζωής ουσιαστικά. Πώς θέλουμε λοιπόν να προωθήσουμε αυτή την ιδέα ε, του δίκαιου ανοιχτού εμπορίου μεταξύ των πολιτών. Θα συνεχίσετε λοιπόν το έργο το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει στην προηγούμενη θητεία. Με τα χαρά, λέει ο κύριος Χόγκαν, να προωθήσω το δίκαιο εμπόριο. Fair and ethical trade. Η Γάνδη πήρε το βραβείο το σχετικό το 19 και βεβαίως και θα στηρίξω και ε, την πρωτοβουλία για τη συνέχιση απονομής αυτού του βραβείου τα επόμενα χρόνια, διότι μπορεί σίγουρα να βοηθήσει τις πληροφορίες που έχουν στη θέση μας να τις διαθέσουμε, να τις αξιοποιήσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να βοηθήσουμε στη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των πολιτών, να κάνουν σωστές αγορές προϊόντων από τις διάφορες χώρες του κόσμου. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, εδώ ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος. Ακούσαμε τους συντονιστές από τις πολιτικές ομάδες. Προ τον υποψήφιο Επιτροπό Φιλ Χόγκαν και έχουμε τώρα 18 ακόμη ομιλητές με βάση το περίφημο σύστημα DEONT. Γιώργεν Βάρμπορν ο πρώτος. Um, Ευχαριστώ. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχω μια ερώτηση που είναι και σπονδυλική στήλη, είναι ραχοκοκαλιά της οικονομίας της Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ηγήθηκε των διαπραγματεύσεων ε, για νέες εμπορικές συμφωνίες ε, με τους περισσότερους ε, από άλλα, εταιρικά, ε, από άλλα μπλοκ, άλλες χώρες. Όμως οι ΜΜΕ πολλές φορές δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που δημιουργούν υποτίθεται για αυτές, αυτές τις νέες εμπορικές συμφωνίες. Μόνο τα δύο τρίτα των εξαγωγιών να χρησιμοποιούν αυτές τις συμφωνίες ελεύθερο εμπορίου. Επομένως, έχω τις εξής δύο ερωτήσεις. Ποια συγκεκριμένα μέτρα θα λάβετε ώστε να αυξήσετε τα ποσοστά αξιοποίηση των FTA των Συμφωνιών Ελεύθερη Πορεία από ΜΜΕ. Και δεύτερον, θα πιέσετε για πιο ευέλικτο και σαφεί κανόνε προέλευση, ώστε οι εξαγωγεί και οι εισαγωγεί να μπορούν να αξιοποιήσουν αυτέ τι εμπορικέ συμφωνίε. Απάντηση. Όπω είπατε, πράγματι υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις, μικρομεσαίες, το 80% όπως είπα 700.000 ε, εξάγουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πάνω από το 1 τρίτο των ε, εξαγωγών εισαγωγών 6 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Είναι ένα πράγματι πολύ σημαντικό κομμάτι τη Ευρωπαϊκή οικονομίας. Ξέρετε, έχουμε πλέον ε, κεφάλαια αποκλειστικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εμπορικέ συμφωνίε. τι μπορούμε να κάνουμε για να τι βοηθήσουμε και πάντοτε σε κάθε νέα συμφωνία θα υπάρχει ένα τέτοιο αποκλειστικό κεφάλαιο για τι ανάγκε του συγκεκριμένου αυτού τομέα, τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Και βέβαια υπήρξε ένα πρόβλημα να ενημερωθούν σωστά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το είπα και σε προηγούμενη απάντησή μου. Το Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη και εμεί, οι αιρετοί έχουμε ένα ρόλο να δραματίσουμε σε κάθε κράτο μέλο, για να μπορέσουμε να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση και να δημιουργήσουμε νέε πλατφόρμες στα κράτη-μέλη ώστε να αναπτυχθούν συγκεκριμένε δράσει για τι μικρομεσαίε αυτέ επιχειρήσει. Βεβαίω και είμαι πρόθυμο να ακούσω ποιε είναι οι βέλτιστε πρακτικές. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα η Κομισιόν, ούτε και η εμπορική πολιτική μπορεί να τα κάνει όλα. Αλλά αν έχουμε μια καλή συμφωνία και είναι κρίμα αν υπάρχει ένα καλό κεφάλαιο στη ΜΜΕ να μην μπορούν να το αξιοποιήσουν οι ΜΜΕ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι αντικείμενο των διαβουλεύσεων και διαπραγματεύσεών μα με του εταίρου οι κανόνε προέλευση. Υπάρχουν σίγουρα ε, προβλήματα πολλέ φορέ και προσπαθούμε να τα μετριάσουμε με τις συμφωνίες μας στο βαθμό του δυνατού. Θέλουμε να είναι συνεκτικοί οι κανόνες προέλευσης στις διάφορες εμπορικές συμφωνίες και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το πετύχουμε. Ένα σημαντικό για όλες τις επιχειρήσεις θέμα και ιδίως για τις μικρομεσαίες βέβαια είναι η γραφειοκρατία. Και γνωρίζω ότι στη, στο Mission Letter θα προσπαθήσετε λέτε να τα πλουστεύσετε one in, one out, ένα προς ένα. Πώς θα την εφαρμόσετε στην πράξη την αρχή αυτή στο τομέα του εμπορίου. Απάντηση. Πρόεδρος Φοντερ Λάιεν στις ε, κατευθυντήριες γραμμές έκαμε πολύ βαρύνουσα δήλωση και σίγουρα ε, υπάρχει ένα πρόβλημα γιατί δεν έχουμε τόσο πολύ νομοθεσία. Θα προσπαθήσουμε να ε, βελτιώσουμε την νομοθεσία και έχω και εγώ το ρόλο μου. Και φαντάζομαι ότι θα βρούμε κάτι. Ε, γιατί πράγματι υπάρχουν αλληλεπικαλύψεις και υπάρχει δικαιωτικό άχθος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα το δούμε αυτό. The next is Nicola Ο επόμενος είναι ο Νικολά Ντάντι. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αν συμφωνείτε, να αρχίσουμε από το θέμα του ΠΟΕ. Κάποιοι συνάδελφοι ήδη το έθιξαν. Πρόκειται για θεσμική πολιτική κρίση στην οποία βρίσκεται γιατί έχουν μπλοκαριστεί οι πολυμερείς σχέσεις και ήδη μας είπατε στην ε, απάντηση ότι ε, οι αρνητικές συνέπειες σας απεισχόλησαν εκεί ε, και επομένω είναι πολύ σημαντικός στόχος του 2020 έω 2022 να βρεθεί κάποια λύση. Οπότε θα ήθελα να μου πείτε με περισσότερες λεπτομέρειες αυτό το οποίο θίξατε, αλλά πέστε μου πιο συγκεκριμένα. Έχουμε τις δύο προτεραιότητα της Επιτροπής για αυτή τη θητεία, την αλλαγή του κλίματος και το κοινωνικό θεματολόγιο. Εσείς πώς θα τα προωθήσετε αυτά στα πλαίσια του ΠΟΕ, Χόγκεν. Όπως είπα προηγουμένως, προσπαθούμε να συνεχθούμε με εταίρους μας που είναι στο ίδιο μήκος κύματος για να μην έχουμε το Δεκέμβριο κατάρρευση των πραγμάτων στο δεύτερο βαθμίο όργανο, ακόμα είπατε να απήντησαν και το θεματολόγιο μας είναι να έχουμε καινούριου κανόνες για να υπάρξει κλίμα δίκαιο για τις επιδοτήσεις, για την τεχνολογία, θα πρέπει να θωρακίσουν περισσότερο το νομικό πλαίσιο. Διαφάνεια επίσης, ε, μεταφορά τεχνολογίας κλπ. Και να δούμε τι θα γίνει με τον ΠΟΕ και την Κίνα. Και επίσης είναι σαφές ότι όπως έχει σήμερα ο ΠΟΕ δεν είναι αποδοτικός και αποτελεσματικός. Είπαμε ότι μίλησα σήμερα με τον Γενικό Διευθυντή. Συμφώνησε. Θα πρέπει η διαδικασία λήψη αποφάσεων να γίνει πιο γρήγορη να δούμε τι γίνεται και με την πολιτική έκθεση. Να σταματήσει να υπάρχει αυτό το απόλυτο μπλοκάρισμα. Επίσης, συζητείτε επίσης το τι θα πει επίπεδο ανάπτυξης χώρας. Μιλούμε για οικονομικές ατμομηχανές της παγκοσμίας οικονομίας. Τέτοιου είδους χώρες εξετάζουμε. Δεν θα πρέπει να υπάρχει δυσμενής διάκριση, προτιμήσεις. Να, τι μεταρρυθμίσεις θέλουμε ε, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Ντάντε. Όχι. Ε, κάνει την επερώτηση τώρα ο Ντάντε. Αλλά δεν ακούγεται. Για να δούμε κάτι άλλο κάτι άλλο, τι είπαμε, τι θα γίνει με τα ψηφιακά, το, το ηλεκτρονικό εμπόριο, όλα αυτά ήδη τα έχουμε θίξει, θα πρέπει να προστατευθούν οι Ευρωπαίοι. Γιατί έχουμε ένα σωρό εμπορεύματα που εισάγονται στην Ευρώπη με την ψηφιακή, μεθοψηφιακή αγορά. Επίσης θα πρέπει να προστατευτούν τα προσωπικά δεδομένα των Ευρωπαίων. Και επίση επ' αυτού θεωρώ ότι θα πρέπει κάτι να κάνουμε μέσω του ΠΟΕ και σε αυτό το μέτωπο. Και εκεί να είμαστε κάθετοι και αποφασιστικοί και εσείς κάτι να κάνετε για την προστασία των Ευρωπαίων για αυτό το τόσο σημαντικό που είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ο υποψήφιος επίτροπος. Δύο είναι οι στόχοι τα δεδομένα και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Θα πρέπει να προστατευτούν τα μεν και να είναι ανοιχτό το δε. Να, τι είδου συνομιλίε γίνονται στον ε, ΠΟΕ και όλο ένα και περισσότερο εξοικειώνομαι για το θέμα, γιατί έχουμε πρόσφατα υποβάλει αναθεωρημένες προτάσεις για να ξεμπλοκάρουμε την κατάσταση, να εκμεταλλευτούμε τα περιθώρια που υπάρχουν και προσδοκάτε περισσότερη πρόοδος των πραγμάτων. Και ελπίζω μέχρι τον Ιούνιο του χρόνου να έχουμε συμφωνήσει κάτι να γίνει με την Κίνα, κάτι να γίνει με η Ιαπωνία και τη ΣΥΠΑ. Να, και αυτή είναι σημαντική παίκτας πέραν ημών. Άρα να δούμε τι θα γίνει με τη τεχνολογία, για τις επιδοτήσεις, για την πνευματική ιδιοκτησία. Πρέπει να προχωρήσουμε σε όλα αυτά τα μέτωπα αν θέλουμε να υπάρχει πρόοδος. Έτσι να υπάρχει η, η ενιαία ψηφιακή αγορά που να ωφελεί τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Να υπάρχει ένα στεγανό πλαίσιο και αυτό να αποδίδει σε παγκόσμια κλίμακα. Ο πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ και ο επόμενος. Τζόρντι Κάνιας. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Χόγκαν, επί τη βάση των εγγράφων σας απαντήσεων είπατε ότι θα κάνετε κάτι για το Μερικοσούρ, αλλά πέστε μας πιο συγκεκριμένα. Πέρα τώρα είπατε και στην εισήγησή σας σε σημαντικούς τομείς. Προσφέρονται έτσι ευκαιρίες και έτσι να δυναμώσει η παρουσία της Ευρώπης σε μια τέτοια συγκυρία που με τις άμεσες επενδύσεις θέλουν να μας υπερκυράσουν οι ανταγωνιστές μας. Τώρα τι θα γίνει, υπάρχουν κάποιου είδου ε, θεμητές επιφυλάξεις ε, από πλευρά γεωργών, από πλευρά κοινοτρόφων και επίσης υπάρχουν κάποιες άλλες ε, θεμητές επιφυλάξεις από άλλους κλάδους, γιατί είδατε τι έγινε με τον Αμαζόνιο, που είναι θέμα των κεφαλαίων για το περιβάλλον. Πέστε μου, τι θα κάνετε ούτω ώστε να υπάρχουν εγγυήσει μια ισότιμη, δίκαιη, ισορροπημένη, ε, βιώσιμη συμφωνία με τον Μερκοσούρ και να υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί ούτω ώστε να μπορούμε να πετύχουμε του περιβαλλοντικού μα στόχου και εν και του τι συμφωνήθηκε στο Παρίσι, αλλά επίση να καλυφθούν και οι εργασιακέ συνθήκε και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ, Χόγκαν. Όπω προείπα, θα ήταν ε, όλο το επιχείρημα για όλα αυτά. Δεν θα, είχαμε, δεν θα είχαμε κανένα είδου ε, μόχλευση, α πούμε, αν δεν υπήρχε η εμπορική συμφωνία. Βεβαίω, καταλαβαίνω σε αυτέ τι επιφυλάξει των ε, ε, ε Γεωργών, εσεί στη χώρα σα θέλετε τη συμφωνία Μερκοσούρ. Νομίζω ότι οι περισσότεροι κλάδοι στη χώρα σα γιατί ωφελούνται πάρα πολύ. Άρα θα ήταν κάτι πάρα πολύ θετικό. Τον υπάρχει ε, αυτή η συμφωνία, να υπάρχει κάποιο είδου απορρίθμιση εμπορική και επίση έτσι θα υπάρχει και προστασία ε, των προϊόντων με ε, γεωγραφική προστασία. Πολλές φορές έχουμε κάποιους αντιπάλους στην παγκόσμια σκηνή που δεν εκτιμούν το ε, τις δικές μας κατακτήσεις από πλευράς προστασίας, προέλευσης κλπ. Οπότε θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη και στη Γεωργία. Έτσι να κάνουμε τη διαχείριση των πραγμάτων. Πρόσβαση στην αγορά όσον αφορά τη διαδικασία επίλυσης ε, διαφορών και αυτό για μας είναι ένα πλεονέκτημα Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει σχέση με τη Συμφωνία των Παρισιών, όπου η Νότιος Αμερική έχει προσχωρήσει και καλύτερα είναι τα πράγματα από ότι να έχει φύγει όπως κάνουν οι Άρα, είναι πάρα πολύ θετικό να προσχωρήσουν σε αυτή την υπόθεση τέσσερις ε, εν λόγω νότιοαμερικανικές χώρες. Άρα πρέπει να σταθμίσουμε τα πράγματα. Αλλά ιδίω όσον αφορά το πλεονέκτημα από την πρόσβαση στην αγορά. Και αυτό που είπατε θα είναι μια θετική κατάρρευση των πραγμάτων. Επερώτηση. Κάνιας. Ναι, εντάξει. Προφανώς και ε, συμφωνώ. Δεν χρειάζεται να με πείσετε. Αλλά το θέμα είναι πώς θα παρακάμψουμε τις θεμητές επιφυλάξεις. Γι' αυτό σας ρωτάω, γιατί τελευταία υπήρξαν κάποιες ενδείξεις ότι δεν υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου, οπότε δεν πετυχαίνουμε αυτά τα οποία συμφωνήσαμε. Δεν τηρούνται τα συμπεφωνημένα. Πού είναι οι ρήτρε διαφύλαξη. Γι' αυτό ανησυχούμε και μιλάμε για πάρα πολύ σημαντικού τομεί και πάρα πολλοί Ευρωπαίοι απαιτούν το να τηρούνται τα συμπεφωνημένα για το περιβάλλον βάσει τη Συμφωνία των Παρασίων και φυσικά και είναι να μην υπάρξει συμφωνία, αλλά θα πρέπει να μπορέσουμε να δούμε τι θα κάνουμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση, να βελτιώσουμε αυτούς τους ε, μηχανισμούς θωράκισης, εφαρμογής και επομένως να πείσετε αυτούς που δεν έχουν πιστεί. Ο Χόγκεν. Αν φέσεις κάποια χώρα Μερκοσούρ ότι δεν θέλει να συνεργαστεί, δεν θέλει να ε, είναι στη Συμφωνία του Παρισίων, δεν θα γίνει τέτοια εμπορική συμφωνία. Δεν είναι ιδιώδης η κατάσταση, αλλά είναι μια επιλογή. Αν δεν υπάρξει πρόοδο στον διάλογο που υπάρχει σε, στη, στην κύρωση της συμφωνίας, τότε έχουμε αυτήν την επιλογή. Και τους το λέμε των εταίρων μας στο Μερκοσούρ. Έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Άρα υπάρχει πίεση μεγάλη και επί αυτών για να εξασφαλιστεί ότι θα υπάρξει για τη διαδικασία της κυρίως της συμφωνίας θετική κατάληξη. Αλλά αυτός ο μηχανισμός της θωράκισης αφορά πρώτα πρώτα γεωργία και για πρώτη φορά υπάρχει τέτοιος μηχανισμός για τα πρόεδρα που μας ενδιαφέρουν. Καμπότζη, Μιανμάρ, από πλευρά Ισπανία, Ιταλία. Έγινε αυτό. Και χωρίς προηγούμενο αποδίδει το σύστημα. Έχουμε τις εγκρίσεις ελέγχουμε το πού γίνεται η αδειοδότηση για το βόλιο, ότι εισάγουμε, να έχει ελεγχθεί 100%, να είναι στα δικά μας πρότυπα. Οπότε θα πρέπει σωστά να έχουν καλύτερη επικοινωνία. Αλλά βεβαίως να υπάρχει σωστή και ακριβή ενημέρωση. Ε, ευχαριστώ. Η κυρία Άννα Μισέλ Σιμακοπούλου. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτρόπε, λέτε στην Επιτροπή σας ότι η Ευρώπη βρίσκεται στην καρδιά του πολυμερού συστήματος. Τι προτεραιότητες έχετε, τι θα γίνει με τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕΙΔΙΟΣ στον τομέα της τεχνολογίας τη μεταφορά τεχνολογία και του ηλεκτρονικού εμπορίου, πώ θα θωρακίσετε την ηγετική θέση τη Ευρώπη και σε σχέση με ΕΠΑ και σε σχέση με Κίνα. Άρα, διπλή ερώτηση σα κάνω πρώτα-πρώτα, πώ θα εξισορροπήσετε ε, αυτέ τι τάσει ε, ελεύθερο εμπόριο, ε, πολυμερέ σύστημα, προστατευτικά συστήματα, άλλα μέσα πολιτική στα πλαίσια του που έχει τα του και δεύτερον. Πώς προτίθεστε εμείς, η Επιτροπή μας, να εμπλαγεί στις προσπάθειές σας για την μεταρρύθμιση του ΠΟΕ. Αυτό το γράψετε στην ε, έγγραφη απαντήσή σας και λέτε ότι είναι προτεραιότητά σας. Χόγκεν, όπως προανέφερα, ο ΠΟΕ τώρα βρίσκεται στη μεγαλύτερη κρίση που έχει περάσει από τότε που συγκροτήθηκε και τα ξέρετε τα προβλήματα, τι γίνεται με τον μηχανισμό διαφορών, τι γίνεται με τους κανόνες για διαφάνεια και εμεί θα συνεχίσουμε να κάνουμε πέρα από το χέρι μας τον ΠΟΕ. Θα προσπαθήσουμε να βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς εμπορίου. Θα πρέπει να προστατεύσουμε αυτή μας την ε, προσέγγιση βάσει των κανόνων που υπάρχουν. Αλλιώς έχουμε τον νόμο της ζούγκλας. Σε μια σειρά ζητημάτων συμφωνούμε με τη ΣΥΠΑ. Αλλά δεν έχουμε ενδείξεις ότι θέλουν να συνεργαστούν με εμά ή με οποιονδήποτε άλλο για τι αναγκαίε μεταρρυθμίσει στον ΠΟΕ. Το ξέρει και ο ίδιο ο ΠΟΕ ότι πρέπει να μεταρρυθμιστεί. Θα πρέπει όμως να προστατεύσουμε και να προτάξουμε τις αξίες, τα συμφέροντα, ε, περισσότερο από όσο σήμερα. Ε, γι' αυτό και έχει σημασία η άμυνα, η εμπορική άμυνα. Οπότε είναι πολύ σημαντικά αυτά τα οποία και σε επιδιώκετε και έχετε πολλή δουλειά μπροστά σας. Οπότε συνεργαστούμε με το Κοινοβούλιο για να, υπάρχει, να υπάρχουν ε, σωστά μέσα πολιτικής για όλα αυτά τα ζητήματα που πρέπει να επιλύσουμε με αφορά τεχνολογίες, ε, πνευματική βιομηχανική ιδιοκτησία, κινέζικες επιδοτήσεις, εισβολή τέλο πάντων της Κίνας σε αγορές όπως στην Ευρώπη, προστασία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ισότητα, στο δικαιοσύνη στο εμπόριο. Έτσι να γίνει το άνοιγμα. Θα πρέπει και άλλοι να το κάνουν αυτό και να τηρήσουν αυτό το οποίο υποσχέθηκαν. Εδώ και πολύ καιρό στον ΠΟΕ. Ρώτησε η κυρία Σιμακοπούλου. Για πες μας με δύο λόγια, τι θέση έχετε σε σχέση με το διεθνές εμπορικό δίκαιο για τις διεθνείς ε, επενδύσεις. Τι θέλετε να κάνετε με το σχετικό όργανο που αφορά τις επενδύσεις. Με δύο λόγια, είναι μια πολύ πρόσφατη πρωτοβουλία, αλλά βεβαίω και θέλουμε να υπάρχει αυτό το πολυμερές δικαιοδοτικό όργανο. Κάνουμε ό,τι χρειάζεται, αλλά ακόμα είμαστε στην αρχή της διαδρομής. Αλλά όντως χρειάζονται τέτοια όργανα για να λάβει σαρακιουστά η εμπορική πολιτική. Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. επόμενος. Πινιέρα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, μιλήσαμε πολύ και συμφωνούμε Μιλήσαμε λοιπόν για την ανάγκη να προωθήσουμε το πολυμερές εμπορικό σύστημα βάσει κανόνων, τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ και αναφερθήκατε και στην απαραίτητη συμμετοχή των ΗΠΑ, αλλά υπάρχει και η Κίνα. Και βέβαια θα πρέπει να έχουμε υπόψη το ότι η Κίνα έχει επωφεληθεί από ένα σύστημα που της επέτρεψε να προωθήσει τελικά τον αθέμητο ανταγωνισμό. Άρα αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη στη μεταρρύθμιση. Πώς λοιπόν η Κίνα θα συμμετέχει, θα αναλάβει τις ευθύνες τη, στο πλαίσιο του, ε, της μεταρρύθμισης του ΠΟΕ και ταυτόχρονα πώς ε, θα επιτύχετε να ενισχύσετε πραγματικά τα μέτρα εμπορική άμυνα ε, και τη ρήτρα διασφάλιση σε κάθε συμφωνία. Θα ήθελα κυρίω να μου πείτε αν θα λάβετε υπόψη το κόστο που συνεπάγεται για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει και του αγρότε μα το ότι πρέπει να φέρουν το βάρο τη απόδειξη από οικονομική και γραφειοκρατική πλευρά. και αν θυμηθώ και το χαρτοφυλάκιο που είχατε, που ήταν η γεωργία. Τι θα κάνετε για να εξασφαλίσετε την καλύτερη προστασία των πιο ευαίσθητων γεωργικών κλάδων. Κοιτάξτε, από την επαφή μου με κάποιους ήδη θεωρώ πως ε, πολλές χώρες ε, θέλουν να ε, φροντίσουν να συνεχιστεί η διαδικασία του που έχουμε συνεργαστεί με τον Καναδά για μια νέα διαδικασία διαιτησίες ενδιάμεση. Βεβαίω ελπίζω να έρθουν και άλλες χώρες γιατί δύο χώρες δεν φτάνουν ούτε καν δύο γεωγραφικές περιοχές για να έχουμε ουσιαστικό αποτέλεσμα. Επίσης ε, θέλω να έρθω σε επαφή και με τις ΗΠΑ να δω το τι θέλουν γιατί δεν μας έχουν πει τι θέλουν Άρα το ότι κάνουμε κάποιες προτάσεις στη ΣΥΠΑ εδώ και μερικούς μήνες. Οπότε, εντάξει, ξέρω ότι μπαίνουμε και σε μια περίοδο προεκλογική της Ιπά που ίσως επηρεάσει την στάση τους, αλλά στην διαδικασία αυτή έχουμε μια επαφή με την Κίνα. Όχι με τις Ιπά αυτή τη στιγμή. Και ελπίζω να αποκτήσουμε. Το κόστος του συστήματος αυτού υποψιάζομαι ότι σκέφτεστε κάποια συγκεκριμένη νομοθεσία που ίσως έχει δραματικό αντίκτυπο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εξαρτάται βέβαια από το που θα καθορίσουν το όριο οι συνομοθέτες. Για το αν δηλαδή θα είναι βαρύ το κόστος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή όχι. Θα δούμε λοιπόν ε, πώς θα είναι η νομοθεσία που θα πάει στον τριμερή διάλογο πρέπει να ορίσουμε το κατόφλι σε ένα λογικό επίπεδο. Το κόστος έχει τεράστια σημασία από την σκοπιά των μικρών επιχειρήσεων και το πώς θα αντιμετωπίσουν αυτό το κόστος. Οπότε αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχετε και άλλη ερώτηση. Και στη γραπτή σας απάντηση για την εμπορική στρατηγική αλλά και στις παρεμβάσεις σας απόψε δεν μιλήσατε για τις οικονομικές εμπορικές ε, σχέσεις και για τη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λατινικής Αμερικής. Δεν είναι προτεραιότητα. Ε, δεν έχετε αναφερθεί καθόλου. Κάτι άλλο που με ανησυχεί είναι Λέτε ότι θέλετε να ληφθεί υπόψη διάσταση του φύλου στις εμπορικές ε, συμφωνίες, αλλά δεν ε, χαρακτηρίστηκε και από τόσο υψηλό επίπεδο φιλοδοξίας ε, η απάντηση που δώσατε. Η Επίτροπος Μάστρομ έχει κάνει πολλά για την συμπερίληψη της διάστασης του φύλου σε εμπορικές συμφωνίες, τη συμμετοχή των γενικών. Εσείς δεσμεύεστε εξίσου και υπάρχουν κάποιοι αλλά υπάρχουν ε, άλλα προβλήματα. Ε, δεν υπάρχουν ε, κυρώσεις ε, παραδείγματος χάρη για παραποιημένα προϊόντα που έρχονται από το Κίνα. Έχουμε γεωργικά προϊόντα ε, που είναι πολύ ελαττωματικά, μπορεί να μην τηρούν τα φυτογενομικά ε, πρότυπα. Ε, οι κυρώσει τα πρόστιμα δεν είναι ομοιογενή. Ε, θα προσπαθήσετε να προωθήσετε μια καλύτερη τελωνιακή ένωση. κανένα προϊόν σήμερα με το σύστημα δεν μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά μόνο υπό την αιγίδα του συστήματος αυτού του SPS και τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για τους ελέγχους. Και όταν είχαμε το σκάνδαλο στη Βασιλεία πριν από 2-3 χρόνια, αυτομάτως είχαμε 100% ελέγχους για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα. Οπότε αν υπάρχουν παράπονα ή στοιχεία για οποιοδήποτε τέτοιο πρόβλημα, πρέπει να το λέτε πρώτα απ' όλα στο κράτος μέλος, που λειτουργεί με βάση τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, είναι πολύ ισχυρό το κεφάλαιο αυτό και δεν είναι διαπραγματεύσιμο στις ε, συμφωνίε. Όλοι πρέπει να έχουν προδιαγραφέ Ευρωπαϊκή Ένωση Για την ισότητα των φίλων χαίρομαι που αναφέρατε αυτά τα οποία είπε η κυρία Μάνστρομ γιατί δικαίω το ανέφερε αυτό σήμερα. Ίσως ήσασταν παρούσα και είμαι σίγουρη βεβαίως ε, πως έχει ένα πρόγραμμα για το τι πρέπει να γίνει ε, στον τομέα της ισότητας. Οι Ιρλανδοί εδώ βουλευτές θα σα πούν ότι δεν έχω πρόβλημα με το να προωθήσω την ισότητα όταν μιλάμε ε, για τη συμμετοχή στις εκλογές. Ε, στη χώρα μου ο Υπουργός ε, Περιβάλλοντος τέτοια νομοθεσία για να μπουν περισσότερες γυναίκες στην πολιτική με καλά αποτελέσματα. Οπότε δεν χρειάζεται να με πείσετε εμένα, σας διαβεβαιώ για τα ζητήματα ισότητας. Και αν ε, βεβαίω θα καταφέρουμε αυτό για να πετύχουμε τους στόχους ε, αυτούς, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Άννα Καβατσίνη έχει τον λόγο. Καλησπέρα κύριε υποψήφιε επίτροπε. Κύριε Χόγκαν, το χαρτοφυλάκιο σας καλύπτει την ε, πολιτική προστασία των επενδύσεων. Ε, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο όμω εκεί πέρα σε αυτό το οποίο μα είπε η κυρία Φοντερ Λάιν. Κάτι το οποίο είναι ατυχέ, γιατί τα τελευταία χρόνια τα ειδικά δικαιώματα των ξένων επενδυτών έχουν αυξηθεί και ανησυχούν του Ευρωπαίου πολιτε. Και τα έργα επίση στον ε, δικό σας τον τομέα είναι πάρα πολλά. Έχουμε την πολυμερή συμφωνία, την επενδυτική συμφωνία με την Κίνα, την ενεργειακή χάρτα και ταυτόχρονα έχουμε υποθέσεις δικαστηρίου κατά της ε, σταδιακής κατάργησης ε, άνθρακα και ορυκτών καυσίμων. Ανισχύτε λοιπόν μήπως ε, επηρεάσουν αυτά την επίτευξη των στόχων μας και κυρίως την μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής και αν ναι θα διασφαλίσετε ότι οι στόχοι αυτοί θα προηγηθούν των δικαιωμάτων των επενδυτών ειδικά σε σχέση με το πολυμερές δικαστήριο. Και τέλος υπάρχουν τα δικαιώματα των επενδυτών. Είστε ικανοποιημένος και σκοπεύετε να επιβάλλετε και υποχρεώσεις των επενδυτών, π.χ. ανθρώπινα δικαιώματα και περιβάλλον. Και υποκλίνομαι εδώ πέρα στις γνώσεις σας γιατί ήσασταν επί πέντε χρόνια υπεύθυνοι του κόμματός σας. Οπότε, εντάξει, παρόλα αυτά είμαι υπέρ ε, της ε, σύστασης του συστήματος αυτού, όπως είχα πει και νωρίτερα. Ε, για κάποιες εταιρείες ε, οι οποίες έχουν κατασταθεί σε άλλες χώρες. Όμως τέτοιοι κανόνες προστασίας των επενδύσεων είναι ενσωματωμένοι και υπάρχουν ε, στο νομικό σύστημα των κρατών μελών. Μπορεί να μην υπάρχει πάντα εγγύηση σε άλλες χώρες και το νόημα είναι ακριβώς να υπάρχει ένα δίκτυο ασφαλείας. Οπωσδήποτε εγώ δεν είμαι ειδικό ε, σε όλα αυτά, αλλά ε, είμαι διατεθειμένος να έρθω σε επαφή μαζί σας για να δούμε το ζήτημα αυτό με τρόπο ουσιαστικό για να δούμε το τι συνέπειες έχει ανεξαρτήτως των όσων είπαμε ότι τα δικαστήρια αυτά είναι σημαντικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω άλλη μία ερώτηση ε, και για αυτό το θέμα και για την ε, για τις ερωτήσεις των συναδελφών γιατί έχουμε το κεφάλαιο του βιώσιμου εμπορίου των στόχων των αναπτυξιακών, γιατί είπατε ότι πρώτα απ' όλα θα αναφερθείτε στην επιβολή και αυτό είναι σωστό. Αλλά αναρωτιέμαι, καθώς οι στόχοι αυτοί είναι καινούργοι και περιλαμβάνονται βεβαίως και στην επιστολή σας, τι νέες προτάσεις έχετε για να εφαρμοστούν και σε όλες, σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες, όχι μόνο στο σχετικό κεφάλαιο. Κοιτάξτε, απάντηση. Ήδη έχουμε τις δεσμεύσει μας ε, για την ε, Συμφωνία των Παρισίων ε, και στους βιώσιμους στόχους, στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Οπωσδήποτε αυτό δεν εμποδίζει τον ΠΟΕ να τα ενσωματώσει. Σε αυτό περιλαμβάνει και πολλές δεσμεύσεις που έχουν προσυπογράψει διάφορες χώρες. Επίσης, μετά την ε, συζήτηση το 2017-18 αναπτύξατε ένα σχέδιο δράση 17 σημείων που αφορά ακριβώς ε, το κεφάλαιο αυτό το οποίο πράγματι θεωρώ ότι είναι μια ατζέντα, ένα πρόγραμμα εργασίας. Και νομίζω λοιπόν ότι το πρόγραμμα αυτό, είτε στον ΠΟΕ, είτε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αν μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτού του στόχου, ε, θα επιτύχει μεγάλη πρόοδο τα επόμενα πέντε χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος ε, Κάμπο Μενόζη. Σας ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε κύριε Επίτροπε. Έχουμε την απόφαση για την Airbus στον ΠΟΕ, μια πολύ ευαίσθητη περίπτωση και βεβαίως μια χώρα η οποία δεν συμμετέχει στο Airbus, η Ιταλία, θα είναι η χώρα η οποία θα έχει το δεύτερο μεγαλύτερο πλήγμα από την εφαρμογή των νέων Αμερικανών, Αμερικανικών δασμών. Και κυρίως ο τομέας της ε, γεωργίας ε, θα πληγεί. Οπότε ελπίζω ότι θα είναι, καταβάλλετε τις ε, κατάλληλες ε, προσπάθειες για να βρεθεί ένα καλύτερο σημείο ισορροπίας όσον αφορά την εφαρμογή της απόφασης αυτής, γιατί βεβαίως το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ήσασταν και Επίτροπος Γεωργίας μέχρι τώρα, πως το Μερκοσούρ Βεβαίω, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, αλλά και όλες αυτές οι χώρες ε, έχουν συμφωνίε που αφορούν πολύ τον ε, ε, γεωργικό τομέα. Φαντάζομαι λοιπόν ότι θα σας απασχολεί το ζήτημα. Κοιτάξτε, η γεωργία δεν είναι τμήμα διαπραγματεύσεων με τη ΣΥΠΑ. Δεύτερον, θα ήθελα είπα, να έρθουν σε επαφή μαζί μας, γιατί η Airbus πρέπει να συμβαστεί με την απόφαση του ΠΟΕ και έτσι πρέπει να γίνει. Και αν διαπραγματευτούμε μαζί τους ε, σε σχέση και με την ε, Boeing δεν θα χρειαστεί να επιβάλλουμε αντίπεινα, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε την έκταση των δασμών αν είναι 5 δισεκατομμύρια, 10 δισεκατομμύρια, 25 δισεκατομμύρια. Οπότε όταν δούμε την έκταση που θα έχουν θα έρθω και εγώ σε επαφή με του ενδιαφερόμενους και στην Επιτροπή αυτή και αλλού να δούμε τι θα κάνουμε για να υψώσουμε το ανάστημά μα ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, να δούμε αν θα το κάνουμε αμέσω. Αλλά βεβαίω πρέπει να λάβουμε και υπόψη τα αντίπεινα που ίσω θα επιβάλλουμε στην περίπτωση τη Boeing. Οπότε εγώ θα ζητούσα από τις ΗΠΑ να διαπραγματευτούν μαζί μας αντί να πάμε σε έναν εμπορικό πόλεμο που θα βλάψει και τις δύο οικονομίες και τους δύο κλάδους ε, στην, στον τομέα της αεροπορίας. Έχετε και άλλη ερώτηση? Χούμπνερ, Μάντελσον, Άστον, Φεραίρο Βάλτνερ, Ντεγκούχτ, Μάλμστρομ, ε, Χόγκαν είναι όλοι οι επίτροποι από το 2004 μέχρι σήμερα που εκπροσωπούν χώρες με διαφορετικά εμπορικά συμφέροντα που επηρεάζουν την ε, Μεσόγειο. Θα ήταν σημαντική νομίζω μια νέα προσέγγιση για να ασχοληθεί λίγο η Κομισιόν για να υπεραυστεί τις γεωγραφικές ενδείξεις ε, και την ε, ε, ποιότητα των προϊόντων. Δεν ξέρω μας, αν μπορείτε να μας εγγυηθείτε κάτι τέτοιο, γιατί βεβαίως ε, έχουμε για νιωστή φορά έναν εκπρόσωπο μιας χώρας που είναι μακριά από όλη αυτήν την συζήτηση και την ανησυχία μας και οφείλει να εκπροσωπήσει ολόκληρη την Ευρώπη σε ένα θέμα πολύ ευαίσθητο. Ε, πρώτα απ' όλα δεν είμαι επίτροπο ακόμα, οπότε όταν με βάζετε με του άλλου, βιάζεστε λίγο. Ε, κοιτάξτε, έχω μια δουλειά να κάνω, ξέρετε, ω επιτροπό να υπερασπιστώ τα συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα επιβάλλουμε δασμού ε, εμεί ε, λόγω τη έρμπα. Οι ΗΠΑ θα το κάνουν. Και ελπίζω η Ιταλική κυβέρνηση να ασκήσει την επιρροή της στους φίλους τη ΕΠΑ που ξέρω ότι έχετε πολλούς, να του πείστε ότι η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτό το οποίο πρέπει να γίνει. Έχουμε λοιπόν καταθέσει διάφορες ε, προτάσεις τον Ιούλιο για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία επικοδομητική. Αντιλαμβάνομαι ότι θα υπάρξουν χώρες όπως ε, η δική μου που θα έχουν μια παρόμοια άποψη με την ε, δική σας στην Ιταλία αλλά πρέπει να υπερασπιστούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οπωσδήποτε πρέπει να υπερασπιστούμε και τα εμπορικά μα συμφέροντα παρά το ότι ίσω να μην είναι εύκολο βραχυπρόθεσμα. Σας ευχαριστώ. Γιάννη Ζάχαραντήλο, επόμενος. Ευχαριστώ πολύ. Πίσω σας είμαι. Ακριβώς πίσω σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να στρέψω την προσοχή σας στην Ασία για μια ακόμη φορά. Με πολύ ρεαλιστικό τρόπο μας περιγράψατε τις σχέσεις με την Κίνα ότι δεν είναι ισορροπημένε και πόρο απέχουν τον ανετέλει. Σίγουρα είναι μια πολύ μεγάλη αγορά, άρα μεγάλη ευκαιρία, αλλά δεν είναι και τόσο καλές οι σχέσει. είναι κάπω ταραχώδεις, υπήρξαν ε, κάποια προβλήματα. Έχουμε τη διαδικασία του screening τώρα που εισαγάγαμε. Θα ήθελα όμως να είστε λίγο πιο συγκεκριμένος ω προς το πώς εσείς θα βοηθήσετε να χαραχθεί αυτόνομη στρατηγική των διαπραγματεύσεων που θα έχουμε την Κίνα τον οποίο θα ηγηθείτε. Να μην γίνει ένα copy-paste, αντιγραφή επικόλυση, δηλαδή της πραγματευτικής τακτικής στον ΗΠΑ. Απάντηση. Όπως γνωρίζετε, έχουμε με την Κίνα αυτή τη στιγμή τις διαπραγματεύσεις σε σχέση με μια επενδυτική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα και είναι και μια πολιτική πλατφόρμα για να διερευνήσουμε και άλλα ζητήματα, όλα αυτά τα οποία έχετε θέσει σήμερα μεταξύ αυτών και κάποια τα συγκεκριμένα βήματα που σας περιέγραψα για τις κρατικές ενισχύσεις, ε, την ξαναγκαστική μεταφορά τεχνολογίας, ε, το ότι δεν έχει ανοίξει την αγορά όσο θα είχε ε, με βάση τις δεσμεύσεις κτλ. Μέχρι το τέλος του 2020 πότε θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, το λέει και η κυρία Φοντερ Λάιεν στην αποστολή μου. Αν δείτε όλα τα άλλα είναι ένα σταθμός και με μεγάλη πρόκληση για μένα να, να πετύχω κάτι τέτοιο. Ξεκινάμε όμως 5 Νοεμβρίου στην Σενχάη το ε, συνάντηση του ΠΟΕ. Θα συναντήσω και όλους τους ανώτατους αξιωματούχους ε, πλην του Προέδρου της Κίνας βέβαια και θα συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα μας ενδιαφέρουν μεταξύ αυτών και τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ και την ε, ολοκλήρωση της Επενδυτικής Συμφωνίας που διαπραγματευόμαστε μέχρι τα τέλη του 20. Ευχαριστώ. Έχετε δεύτερη ερώτηση, ναι. Η Κίνα, λέει ο κ. Σαχράντιλ, δραστηριοποιείται σε πολλές άλλες νοτατολικές χώρες νοτατολικής Ασίας. Και πρέπει σίγουρα να υπάρχει κάποια γεωγραφική ισορροπία απέναντι σε αυτή την κινέζικη επιρροή. Πώς βλέπετε εσείς τις ε, σχέσεις χάρη με τις χώρες ΑΣΕΑΝ. Θα πρέπει να συνεχίσουν η προσέγγιση αναχώρα ή θα ήσασταν ε, της άποψης να κάνουμε κάτι ανάλογο με τις χώρες Μερικοσούρ. Δηλαδή μια πιο ε, ευρεία συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΣΕΑΝ απάντηση. Έχει κάνει κάθε προσπάθεια η κυρία Μάλστρομ για αναπεριφέρεια ε, συμφωνίες, όπως παραδείγματος και με τις χώρες ΑΣΕΑΝ. Αλλά υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Ε, είχαμε παραδείγματος ένα πρόβλημα με τις Φιλιππίνες ε, που για τα γνωστά για εσά από το 2015 δεν μπορεί να διαπραγματευτεί. Η Ταϊλάνδη και η Μαλαισία έχουν δυσκολίες σε σχέση και με την εντολή τη διαπραγματευτική που έχουμε για σημαντικά κεφάλαια όπως είναι τα κεφάλαια της μα ανάπτυξης του εμπορίου. Δεν συμμορφούνται Έχουμε όμως πολύ καλή συμφωνία. Παραδείγματος με το Βιετνάμ. Ξέρω ότι η Επιτροπή σας ε, ασχολείται με την φάση της κύρωσης αυτής της συμφωνίας. Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον και ελπίζω να κυρωθεί αυτή η συμφωνία. Και σίγουρα χρειάζονται διευκρινήσεις ε, σε διάφορα ζητήματα. Όταν επισκεφθείτε το Βιετνάμ στα τέλη Οκτωβρίου, ελπίζω να τσέχετε αυτές τις διευκρινήσεις. Επίσης, Σιγκαπούρη. Περιμένουμε να τεθεί σε ισχύ λόγω συμφωνία μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους. Υπήρχαν κάποια ζητήματα, όπως παραδείγματος χάρη οι γεωγραφικές ενδείξεις, αλλά τα λύσαμε. Και βέβαια έχουμε και τη συμφωνία με την Νότια Κορέα από το 2009. Άρα, αναχώρα κάνουμε πρόοδο. Η Ινδονησία έχει μια ευκαιρία, αλλά υπάρχουν δυνατότητες, αλλά υπάρχουν και εκεί προβλήματα, βιωσιμότητα, περιβάλλον. Έχουμε κάνει σημαντικές προτάσει και περιμένουμε την απάντησή τους. Ε, Μπορεί να μην υπάρχει λοιπόν πρόοδος με την προσέγγιση αναπεριφέρεια, αναπεριοχή, αλλά αναχώρα έχουμε πρόοδο. Πρώτος, ευχαριστώ πολύ. Μα ε, κάλυστερο αγαπητός συμπρόεδρος και φίλος είναι επόμενος. Ευχαριστώ κύριε Υποψήφια Επίτροπε. Και η πρόεδρος Φοντριλάιν σας ζήτησε να ενισχύσετε τη δυνατότητα της Ευρώπης να προστατεύει προστατεύεται από αθέμητες εμπορικές πρακτικές μεταξύ άλλων με την χρήση ενός νέου ε, συστήματος για τη διαλογή των ξενάουσων επενδύσεων, το screening που φαίνεται όμως ότι θα συντονίζει στα 12 μόνο κράτη-μέλη ε, την κατάσταση γιατί εκεί υπάρχει αντίστοιχο screening ε, θα τον αναβαθμίσετε αυτό το μηχανισμό για την εξέταση των ξένων επενδύσεων. Ναι, είναι η σύντομη απάντηση. Σίγουρα θέλουμε συντονισμένη, αρμοσμένη προσέγγιση για όλα τα κράτη-μέλη τη Ένωση και ελπίζω να το πετύχουμε. Έχουμε για κάποια κράτη κάποιε ανησυχίε, ιδίω από του φίλου 17 ε, συν 1. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε μία ενιαία θέση ως Ευρωπαϊκή Ένωση για την αναβάθμιση αυτού του μηχανισμού screening που είναι πολύ σημαντικό για να προστατεύσουμε κρίσιμες υποδομές και και συστήματα που έχουμε. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε στην τύχη. Θέλουμε να είμαστε μια ανοιχτή οικονομία. Είμαστε ίσω η πιο ανοιχτή εσωτερική αγορά. Αλλά θέλουμε από του εμπορικού μα εταίρου αντίστοιχα. Η Κίνα μα έχει υποσχεθεί πολλά και δεν τα έχει πραγματοποιήσει μέχρι τώρα. Να δούμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να σημειώσουμε ίσω πρόοδο και στο πλαίσιο τη επενδυτική συμφωνία. Σίγουρα υπάρχουν και άλλα εργαλεία. Παραδείγματο χάρη αυτό για τι διεθνεί προμήθειε που το ξέρετε. Έχετε περώτηση. Ευχαριστώ, κύριε υποψήφιο επίτροπο. Οι παγκόσμιε αγορέ προμηθειών χαρακτηρίζονται από έντονε ανισορροπίε. Είναι ανοιχτή για τρίτε χώρε η ευρωπαϊκή αγορά προμηθειών, αλλά είπατε ότι ε, οι υποψήφοι έχουν να αντιμετωπίσουν ε, τον ανταγωνισμό. Πώς θα το προχωρήσετε αυτό το μέσο λοιπόν ε, των επενδύσεων. Απάντηση. Έχω ξεκινήσει με τον ε, Γερμανό Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Αλτμάιερ, κάποιε επαφέ και το ίδιο θα έχω και τι επόμενε εβδομάδε, εφόσον βέβαια και εκλεγώ. Θα έχω ακόμα περισσότερε επαφέ με Γαλλία και άλλε χώρε για να δούμε ποια είναι τα προβλήματα, ποιοι είναι οι σκόπελοι για μια τέτοια ε, πρωτοβουλία. Είναι σημαντικό να υπάρχουν ισχυρά μέσα εμπορική άμυνα για να διαπραγματευτούμε ορισμένα από αυτά τα ζητήματα που θέλουμε να διαπραγματευτούμε και αντιμετωπίζουμε δυσκολίε προ το παρόν. Πρέπει να έχουμε θέση ισχύω, γιατί έτσι μπορούμε να ασκήσουμε μεγαλύτερη μόχλευση. Σα ευχαριστώ πολύ. Μαριπιέρ Βεντρέν είναι η επόμενη. Υπόψηφε Επίτροπε, είπατε κι εσεί ότι η εμπορική μας πολιτική πρέπει να βασίζεται στην αμοιβαιότητα και σε κανόνισό ισότιμου ανταγωνισμού για να προσπίσουμε τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Πάνω από το μισό των προμηθειών είναι κλειστέ αυτή τη στιγμή ε, λόγω προστατευτικών μέτρων στον ελεύθερο ανταγωνισμό. Συγκεκριμένα λοιπόν, εσεί πώ θα συνεισφέρετε στην απεμπλοκή για τον κανονισμό για την πρόσβαση στις δημόσιε προμήθειε, τι νέε νομοθετικέ προτάσει θα καταθέσετε συγκεκριμένα για να προασπίσετε το πολυμέρε σύστημα και τον σημαντικό ρόλο της Ένωσης. Και σε ό,τι αφορά το σεβασμό της εμπορικής πολιτικής και της εφαρμογής της και ιδίως σε πτυχή της βιώσιμης ανάπτυξης. Είπατε για αυτόν τον chief officer, καλό είναι αυτό, αλλά τι θα κάνει ακριβώς ε, από τη θέση αυτή και επίσης έχετε υποψηφίους και τι δυναμικό, τι ε, ανθρώπινο δυναμικό και τι σχέση με εσάς θα έχει ο, αυτός ο νέος ε, αξιωματούχος. Uh, αν θέλετε να υιοθετήσετε αυτή την, ε, αυτούς τους κανόνες των δίκαιων των ε, θεμητό ανταγωνισμό, σίγουρα πρέπει να ξεκινήσουμε από τον ΠΟΕ, που είναι ο πυρήνας. Εξήγησα στον κύριο Ντάντι, ε, του έδωσα κάποιες ιδέες μου και είπα πώς βλέπω να το πετυχαίνουμε αυτό. Αλλά αν δεν μας υποστηρίξουν οι θα πρέπει να έχουμε ένα εναλλακτικό σχέδιο. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δείξει ηγετική στάση. Το δεύτερο ήμιση του 20 θα το συζητήσουμε την Επιτροπή σας. Τι θα κάνουμε δηλαδή ώστε να υπάρχει ε, και μια διαδικασία επίλυσης διαφορών βάσει κανόνα στα τέλη του 2020. Μίλησα για τα ζητήματα των μέτρων εμπορική άμυνα. Μίλησατε για τι προμήθειε εσεί. Ναι, θέλω να το προχωρήσω και ελπίζω και το Συμβούλιο να αντιληφθεί ότι πρέπει να έχουμε ισχυρά μέσα εμπορική άμυνα στι διεθνεί μα σχέσει για να μπορούμε να διαπραγματευόμαστε με χώρε που δεν παίζουν σύμφωνα με του κανόνε ακριβώ σε σχέση με τι επιδοτήσει ή τη μεταφορά τεχνολογία. Ο Chief Trade Enforcement Officer είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία Τη χώρα σας, ε, στη χώρα σας είναι γνωστό νομίζω και είναι αναπληρωτής γενικός διευθυντής ε, στη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Trade ε, θα είναι και επομένως θα έχει κάποια δύναμη στα χέρια του, στα χέρια της και θα γίνει τέτοια αναδιάρθρωση στην Καμάλτα Τρέντ ώστε να μπορεί με πολύ σημαντικό τρόπο να ενεργεί. Θα του δώσουμε λοιπόν και ανθρώπινο δυναμικό και άλλους πόρους. Δεν θα είναι μια αυτόνομη ε, υπηρεσία. Θα λογοδοτήσει όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Και ελπίζουμε να είναι στο πιο αποτελεσματικός αυτός ε, ο νέος αξιωματούχος. Επερώτηση. Οι Ευρωπαίοι παραγωγοί και καταναλωτέ θα ήθελαν στι εμπορικέ μα διαπραγματεύσει και στι εμπορικέ μα συμφωνίε να έχουμε τι φυτογενομικέ, κοινωνικέ, περιβαλλοντικέ απαιτήσει σε αρκετά εξέχον ε, βαθμό. Συγκεκριμένα τι θα κάνετε για τα εισαγόμενα προϊόντα που μπαίνουν ε, στις ευρωπαϊκές αγορές ώστε να σέβονται πραγματικά τα δικά μας πρότυπα. Απάντηση. Το καλύτερο παράδειγμα που μπορώ να σας δώσω είναι προϊόντα τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο απάτης πρόσφατα. Στο τομέα της Βελογικής Γεωργίας, για παράδειγμα, είχαμε απάτες. Και μεταρρυθμίσαμε τη σχετική νομοθεσία με τη βοήθεια του εισηγητού, Μάρτιν Χάουσλινγκ και την Επιτροπή Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης. Συνεργαστήκαμε στενά, είχαμε μια πολύ καλή ε, τυποποίηση, εναρμόνιση για τους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων τα πρότυπά μα, ε, ε, δηλαδή να γίνονται σεβαστά, να είναι παρόμοια με αυτούς οι οποίοι εξάγουν προς τα εμάς. Και το κεφάλαιο για τα SPS στις ε, εμπορικές συμφωνίες για τα αυτοπροστατευτικά μέτρα. Είναι κάτι που θέλουμε να το καθιερώσουμε σε όλες τις συμφωνίες και θέλουμε να βρούμε μιμητές και σε άλλες χώρες. Θα δούμε τι κάνουμε και με το Αμένο Βασίλειο, αν χρειάζεται να διαπραγματευτούμε. Αν δεν έχουμε τα ίδια πρότυπα, σε αυτή τη γεωργία, βιομηχανικά προϊόντα, αν δεν είναι υψηλά αυτά τα πρότυπα, τότε και άλλες χώρες θα μπορούν ίσως να φέρουν φθηνά τρόφιμα και άλλα γεωργικά προϊόντα σε γειτονικέ χώρες και αυτό θα πλήξει τους δικούς μας παραγωγούς. Θα είναι άδικο και γι' αυτό πρέπει να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα. Ευχαριστώ πολύ, Τιτσιάνα. Λοιπόν. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστούμε κυρία Υποψήφια Επίτροπε. Θέλω να επανέλθω στο θέμα της αξιολόγησης των βιώσιμων επιπτώσεων. Δεν ήταν στο παρελθόν αυτό μια προτεραιότητα, παρά το ότι προφανώς είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν έγινε το ζήγισμα του περιβαλλοντικού και κοινωνικού επιπτυχίου. Ε, βέβαια και ξεκίνησαν ε, πριν γίνουν αυτές οι μελέτες, ε, οι διαπραγματεύσεις και σας ερωτώ εσείς θα αναλάβετε να ολοκληρώσετε τέτοιες μελέτες και να τις δημοσιοποιήσετε πριν αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για τις μέλους συμφωνίες. We uh, Ναι. Κάνουμε τέτοιου είδους μελέτες επιπτώσεων πριν τις διαπραγματεύσεις και τώρα πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για τη βιωσιμότητα, για άρευνα αγοράζει για τις ευκαιρίε που παρουσιάζονται. Και έχουν δημοσιοποιηθεί συμφωνίε σε σχέση με μελέτε σχέση με τι συμφωνίε, μάλλον και η σχετική ε, μελέτη πρόκειται πριν την ακύρωση τη συμφωνία να δημοσιευθεί. Οπότε θα υπάρχει και μια τέτοια μελέτη επιπτώσεων σε σχέση με τη συμφωνία με τις χώρες Μερκοσούρ, να γίνει οικονομική ανάλυση, να γίνει ανάλυση των επιπτώσεων και κατόπιν θα υπάρχει και μια εκ των προτέρων μελέτη των επιπτώσεων. Ε, όπως είχε γίνει πριν από 3-4 χρόνια πριν υπάρξει η εφαρμογή των συνθήκων. Οπότε, όσον αφορά τι αξιολογήσει, δεν μα λείπουν. Και με μεγάλη μου χαρά να κάνω αυτό που είπατε για τη δημοσίευση. Σα ευχαριστώ για την ε, απάντηση. Πριν τι διαπραγματεύσει, λέω όμω, όχι πριν την ακύρωση τη συμφωνία. Και τώρα ε, σκέφτομαι ότι άρα είναι να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσει α πούμε, με κάποιε χώρε που υπάγονται τώρα στο πρόγραμμα ΕΔΙΑ, γιατί είναι το θέμα της εργασίας των ανηλίκων και άλλα θέματα και σε σχέση με αυτό. Μου έρχεται στο μυαλό ένα άλλο θέμα που αφορά την εργοποίηση της ρήτρας διαφύλαξης που ε, ε, επιστάδευσε η Επιτροπή για την Καμπότζη προσέφηκε για αυτό η Καμπότζη και είπε ότι δεν είναι βάσιμο το επιχείρημα για ε, συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ρήτρα μα δεν θα πρέπει να υπάρχει ένας ορισμός για το συμφέρον της Ένωσης ούτως ώστε να μπορεί κανείς να επιστατεύσει, να ενεργοποιήσει αυτή τη ρήτρα ακόμα και να χρειάζεται μόνο ένα κράτος μέλος. Ναι. Τι να σας πω δεν ξέρω να σας πω κάτι για τον ορισμό του συμφέροντος της Ένωσης, αλλά μπορώ να σας πω ότι έχουμε το Everything But Arms ε, σε σχέση με την Καμπότζη, την Μιανμάρ, ε, για το ρύζι, για τις εξαγωγές ε, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιστρατεύσαμε αυτή τη ρήτρα και τελικά βρέθηκαν όλα τα στοιχεία από Ιταλία και Ισπανία, ιδίω από την Ιταλία, ότι υπήρχε μια κάθε απότομη άνοδο των εισαγωγών σε σύντομο διάστημα. Αναλάβαμε ενέργειες, ίσως αργήσαμε λιγάκι, αλλά τα καταφέραμε και για πρώτη φορά επικαλεστήκαμε την ρήτρα διαφύλαξης υπέρ των προαγωγών των χωρών αυτών Ιταλίας Ισπανίας για να τους προστατεύσουμε. Ακριβώς όπως και συμφωνείτε. Και αυτό το αποτελεί προηγούμενο, ούτως ώστε να επικαλεστούμε τη ρήτρα και για άλλα προϊόντα. Μέχρι τώρα είχαμε να κάνουμε με αγορές υπό απορρίθμιση, αλλά τώρα με αυτό το προηγούμενο μπορούμε να το κάνουμε με κάποιο είδους ποσοστώσεις, ε, με δασμολογήσεις ε, που, που κάποια προϊόντα με οποιαδήποτε χώρα στον ε, κόσμο. Να, έγινε αυτό με την Καμπότζη για να προστατεύουν τους όριζο, Ιταλούς και Ισπανούς. Να, επομένως, η Μιανμάρ αποτελεί ένα καλό παράδειγμα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. κύριε Σούστος. Κύριε Χόγγεν, η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν μίλησε για έναν ε, φόρο διοξιδίου του άνθρακα στα σύνορα. Κάτι το οποίο θα επιτρέψει να έχουμε φιλόδοξου στόχου για το κλίμα, αλλά και ταυτόχρονα δικαιού όδου ανταγωνισμού μεταξύ ε, παραγωγών Ευρωπαίων και μη. Θα πρέπει λοιπόν τους επόμενους μήνες να ληφθούν σοβαρές αποφάσεις. Πρώτα απ' όλα να επιλεγεί η νομική βάση, αν θα είναι η περιβαλλοντική ή εμπορική νομοθεσία. Βεβαίως ε, ο φόρος ο οποίος έχει το μειονέκτημα ότι θα πρέπει να εγκριθεί ομόφωνα από το Συμβούλιο Σημαντικό είναι βεβαίως το πώς θα υπολογιστεί και το τι σχέση θα έχει με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών, γιατί θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τον ΠΟΕ και μετά βεβαίως υπάρχει το ερώτημα του αν υπάρχει σχέση μεταξύ του ύψους ε, αυτής της αντισταθμιστικής ε, πληρωμής με την βλάβη στο περιβάλλον. Οπότε το ερώτημα είναι, ε, με βάση αυτά και άλλες ε, πτυχές μπορείτε να μας πείτε ποιο είναι το δικό σας ε, το σχέδιο για τον φόρο αυτό για το διοξείδιο του άνθρακα στα σύνορα. Κοιτάξτε, είναι ένα περίπλοκο ζήτημα και χαίρομαι ιδιαιτέρως για το ότι ο αρμόδιος επίτροπος θα είναι ο κύριος Τζεντιλόνι γιατί αυτός θα ασχοληθεί με όλη τη δύο επιμέλεια με αυτό το ζήτημα και την αξιολόγηση αντικτύπου γιατί είναι ένα περίπλοκο ζήτημα όπως μόλις είπατε και ο στόχος είναι να αποφευχθεί η λεγόμενη διαρροή του άνθρακα και να μπορούν οι εταιρείε να λειτουργήσουν με ίσους όρους ανταγωνισμού και βεβαίως αν συνδυαστεί με δωρεάν άδειε στο σύστημα εμπορία εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε δεν υπάρχει περαιτέρω κόστος. Νομίζω λοιπόν πως αυτή η προσέγγιση, και πρέπει να συνεργαστούμε και με τον Επίτροπο Τίμερμανς, τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο αρμόδιο για τα κλιματικά. Οπότε η εμπορική πολιτική και η μπλοκή της είναι κάτι το θα πρέπει να δω σε επαφές με τους κυρίους Τίμερμανς και Τζεντιλόνι. Προφανώς δεν έχουν υπάρξει συναντήσεις ακόμα, δεν θα υποθέσω εγώ ποιες θα είναι οι θέσεις των άλλων επιτρόπων, θα δούμε ποιε θα είναι οι επιλογέ και θα τι εξετάσουμε προσεκτικά. Δεν θέλουμε να έχουμε μια κατάσταση που εμεί κάνουμε όλα όσα πρέπει να κάνουμε και οι ανταγωνιστέ μα ανά τον κόσμο δεν κάνουν τίποτα. Πώ θα διαχειριστούμε λοιπόν αυτήν την σχέση για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα και ταυτόχρονα ε, οι άλλοι να μην κάνουν ε, τίποτα. Αυτό ε, σημαίνει ότι θα έχουμε ένα ανταγωνιστικό μειονέκτημα. Αυτά θα πρέπει να τα δούμε λοιπόν με μια αξιολόγηση αντικτύπου. Έχετε και περώτηση. Ναι, δεν ήταν πολύ ικανοποιητική η απάντηση, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το να είναι σύμφωνα όλα αυτά με τον ΠΟΕ. Αλλά μια που αναφερθήκατε στο πώς ακριβώς θα μπορέσουμε να επιβάλλουμε τα κεφάλαια αυτά Αναφερθήκατε και στην ε, Νότια Κορέα, όπου ε, υπάρχει ένα πολύ προχωρημένο τέτοιο κεφάλαιο, αλλά πολύ απλά αγνοείται εδώ και 7 χρόνια. Μία. Είμαστε στις συζητήσεις, αλλά στην πραγματικότητα δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Οπότε το ερώτημα είναι πώς τελικά εσείς ως ο αρμόδιος επίτροπος ε, θα επιβάλλετε την εφαρμογή αυτού του κεφαλαίου. Παραδείγματο χάρη να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα περί συνδικαλισμού, κάτι το οποίο προφανώς δεν συμβαίνει στην Νότια Κορέα. Κοιτάξτε, ακριβώς γι' αυτό τον λόγο έχουμε ένα μηχανισμό επίλυσης ε, διαφορών στην Νότια Κορέα για πρώτη φορά σε Συμφωνία ελευθερίου Μπορείου είχαμε μια τέτοια διάταξη. Τώρα πλέον ε, την επικαλείται η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από πολλές προσπάθειες για να υπάρξει ένα σχέδιο δράσης ε, για να ε, τηρήσει αυτό το κεφάλαιο Νότια Χώρα. Οπότε πάμε στο επόμενο βήμα. Ένα μηχανισμό επίλυσης διαφορών με βάση τα συμφωνηθέντα. Τώρα μου λέτε να σας πω ποια θα είναι τα αποτελέσματα σε σχέση με κάτι για το οποίο δεν έχω καμία ιδέα. Ε, και δεν είναι άμεση ευθύνη μου. Και ευχαρίστω βεβαίω να έρθω σε επαφή μαζί σα όταν θα έχω περισσότερε πληροφορίε από τον αρμόδιο επίτροπο ή υπό την ηγεσία του αντιπρόεδρου Τίμερμαν. Ε, εγώ είμαι υπέρ βεβαίω σε ε, διάταξη αυτή, όπω αναφέρω και στην επιστολή μου, να κάνω αυτό το οποίο μου αναλογεί. Αλλά λυπούμε που δεν μπορώ να σα δώσω περισσότερε λεπτομέρειε αυτή τη στιγμή. Δεν μπορείτε ταυτόχρονα να σα δώσω λεπτομέρειε για κάτι το οποίο δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Υπάρχουν ε, περίπλοκα ζητήματα, το γνωρίζετε και εσείς ήδη. Σας ευχαριστώ. Ντανούτα Μαρία Χύπνερ κατόπιν. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας ρωτήσω για το Brexit. Ε, δεν ε, θέλετε να κάνετε εικασίες, αλλά νομίζω ότι αν υπάρξει έξοδος χωρίς συμφωνία, η έφτακτη έξω, ε, δεν θα είναι αυτό το τέλος. Ε, μάλλον αμέσως θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική σχέση και οπωσδήποτε μια συμφωνία ελευθερου θα είναι ο πυρήνας των σχέσεων αυτών. Στο πλαίσιο αυτό γνωρίζω ότι οι Βρετανοί φίλοι μας θα αποφασίσουν τι είδους συμφωνία θέλουν. Γνωρίζω πως η κυρία Μέη ήθελε φιλόδοξες ε, συμφωνίες για μέτρα που θα διασφαλίσουν ε, ένα, ή ένα θα η θα εξασφαλισουν ισως ορους κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερος. Ε, Λαμβάνοντα υπόψη λοιπόν το μέγεθος και την εγκύτητα αυτής της αγοράς, νομίζω ότι οποιαδήποτε συμφωνία εμπορίου θα πρέπει να περιλαμβάνει κάποιες εγγυήσεις και το ερώτημά μου είναι το εξής. Πώς βλέπετε το θέμα αυτών των μέτρων από την σκοπιά των κόκκινων γραμμών για εμάς, ειδικά αν λάβουμε υπόψη την ερμηνεία από την βρετανική πλευρά ότι θα πάνε προς μια ρυθμιστική απόκληση αντί για σύγκληση. Είναι δύσκολο να ξέρουμε ποια κατεύθυνση θα πάρει το ΕΒ Βασίλειο γιατί δεν φαίνεται να συμφωνούν στην Βουλή των Κοινοτήτων όπως επισημάνατε, η Πρωθυπουργό κυρία Μέη και η Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν μια καλή και ισορροπημένη συμφωνία και οπωσδήποτε διαβεβαίωσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση για ζητήματα κρατικών ισχύσεων, δικαιωμάτων εργαζομένων, προστασία των καναλτών, ποιότητα τροφίμων, όλα αυτά που είναι πάρα πολύ σημαντικά και θα παίξουν ένα ρόλο στην εντολή, υποθέτω, που τελικά θα μου δοθεί για να διαπραγματευτώ αυτήν την συμφωνία. Οπότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα έχουν πολλά να πούν στην εντολή που θα δοθεί στην Κομισιόν για να διαπραγματευτεί και είμαι σίγουρος βεβαίω πως ε, θα περιλαμβάνεται εκεί και θα περιλαμβάνονται και οι σύγουροι Σας ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο Μανουέλ Μορέλ. Καλησπέρα κύριε υποψήφι Επίτροπη. Η μεταρρύθμιση στον ΠΟΕ είναι ε, στόχο τώρα η πρόκληση για την εμπορική πολιτική μα. Είπατε για αναγκαστική μεταφορά τεχνολογία, για κρατικέ ενισχύσει, για τον μηχανισμό επίλυση διαφορών, για τι ε, είπα, για πες μας τι γίνεται με την κλοπή πνευματικής ιδιοκτησία, γιατί δεν το είδαμε αυτό ε, στην επιστολή. Τι γίνεται με την παραποίηση, είναι καταστροφή για την Ευρώπη. Αυτό είναι ε, ε, ε, θάνατος για τις ΜΜΕ. Έχουν χαθεί πάνω από 300.000 θέσεις εργασίας. 85 δις ευρώ. Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία πλήσονται. Κλωστεφαντουργία, έπιπλα, φάρμακα, πνευματική Βιομηχανία του και ε, η κυρία Φοντερ Λάιν ε, σιώπησε γι' αυτό. Και για πετε μας, είναι η τη της Επιτροπής. Έχετε έρθει με του ε, Κινέζους γιατί αυτοί απο, ε, εκπρόσωπουν το 80% τη παραποίηση. Τι γίνεται με το Alibaba και το Amazon. Αυτοί πουλάνε προϊόντα ε, παραποιημένα και μίσεις. Τι κάνουμε εμείς, τίποτα. Πρώτα-πρώτα ε, έχουμε προτάξει στους Κινέζους τα μέτρα εμπορικής άμυνας. Έχουν προσφύγει στον ΠΟΕ, έστω και αν έχει κολλήσει το θέμα. Τρίτον, διαπραγματευόμαστε με την Κίνα σε σχέση με επενδύσεις και όλα αυτά είναι υποσυζήτηση. Είναι προτεραιότητα και δική μου και της Κομισιόν. Για να κλείσουμε το 2020 συμφωνία, όλα αυτά που είπατε θα πρέπει να έχουν επιληθεί. Ε, βέβαια, θα τα παρακολουθήσω όλα αυτά από κοντά. Όλα είπα, όσα είπατε. Ναι, είναι αυτός το χαρτοφυλακείο μου, πρέπει να το έχω λύσει μέχρι το 20. l'Europe Ας είναι λιγότερο ωφελές μέχρι τώρα. Η, Ευρώπη μιλούμε για τον ΠΟΕ και λέμε τι ωραία, προχωρούμε τη μεταρρύθμιση τον Ιούνιο, όμως η η Βραζιλία, η Αυστραλία και οι χώρες Μερκοσούρ μας επιτέθηκαν και κατήγγυλαν αυτή την ε, ρήτρα διαφύλαξης, κάτι το οποίο είναι θεμελιώδες για μας. Γιατί το λέω ο συνάδελφός σας, ο κύριος Σεύκοβιτς, που έχει χαρτοφυλακή των προοπτικών, είπε ότι θέλει οπωσδήποτε να στηρίξει τις πολιτικές επί τη βάση κραδάντων στοιχείων και όχι υπό τη βάση ισχυρισμών και ε, ιδεών. Εσείς τι λέτε για την αρχή της διαφύλαξης, τη ρήτρα της διαφύλαξης Πώς τη βλέπετε στα πλαίσια των συμφωνιών ελευθερών εμπορίου. Ήδη φάνηκε αυτό με τη συμφωνία Μερκοσούρ. Εκεί ε, σε αυτή την αρχή. Θα έπρεπε να καλυφθεί από την συμφωνία. Και είδατε τι κάναμε και με την Βραζιλία. Δεν θέλανε, τους πείσαμε. Η για μας ήταν κόκκινη γραμμή. Δεν θα υπήρχε συμφωνία νομίζω εάν δεν υπήρχε η σχετική διάταξη και στη Γεωργία και στα υπόλοιπα. Φέτο φέτος το πετύχαμε αυτό που λέτε. Thanks a lot. ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τζουτ Κέρτον darling Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εσείς, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να πω να για τον Brexit, αλλά και δεν θα το κάνω. Οπότε θα ήθελα να μου πείτε περισσότερες λεπτομέρειες το σύστημα γεννημένων προτιμήσεων είναι ό,τι πιο γενναιόδρο υπάρχει στον κόσμο και αυτό έχει βοηθήσει ευημερία σε πολλές χώρες και περιοχές. Όμως το σύστημα επίσης έχει πολλές τρύπες. Το φάνηκε αυτό από το TST για τις διαφορές Μιανμάρ και Καμπότζια παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα συστηματικά και παραβιάζουν, καταπατούν τις συμφωνίες. Έχουμε τη συμφωνία ε, με προτιμήσεις με τις Φιλιππίνες, γενικέ προτιμήσεις συν και τίποτα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε το σύστημά μα είναι αργό ή αναποτελεσματικό. Τι γίνεται με, το, με την ανάπτυξη, της ρήτρας ανάπτυξης Συμφωνία Ελευθερών Μπορείου. Πέστε μας πέντε πράγματα τα οποία εσείς κάνετε τόσο ώστε να βελτιώσετε την κατάσταση ε, για αποτελεσματικότητα των γενικμένων προτιμήσεων, τόσο ώστε αυτό το, αυτό το μέσο να είναι αποτελεσματικό. Ναι, πρώτα πρώτα έχουμε αυτόν τον Trade Enforcement Officer, τόσο ώστε να επιτηρεί την υλοποίηση αυτών των συμφωνιών παντού. Επίσης, δεχόμαστε καταγγελίες από την κοινωνία, όπως έγινε με το Περού, όπως έγινε με τη διαδικασία διαφορών. η μεθοδολογία name and shame, κατονομασία, καταλογισμός και οπότε νομίζω ότι προχωράνε τα πράγματα σε σχέση με τις συμφωνίες τρίτων. Θέλουμε να εμπλακεί η συμφωνία, η κοινωνία, συγγνώμη, περισσότερε αυτέ αυτές συμφωνίε να υπάρχουν οι πόροι, ούτω ώστε η κοινωνία, η ΜΚΟ, να έχουν τα μέσα για να εμπλακούν. επίση. έχουμε ένα σύστημα εποπτείας για τι γενικευμένε προτιμήσει τόσο ώστε να είναι οι επενδύσει με υπεύθυνο τρόπο, να μην αποτελούν ε, dumping όπως πολλές φορές λέμε και κατηγορούμε άλλους ότι το κάνουν. Επίσης θεωρώ ότι εργασιακά, περιβαλλοντικά είναι θέματα των συμφωνιών που πιστεύω θα τύχουν προτίμησης για τις χώρες γενικευμένων προτιμήσεων, οπότε αυτές οι χώρες θα προχωρήσουν στην εφαρμογή των όσων συμφώνησαν ότι θα κάνουν. συμφωνήσαμε το 2018 και η Επιτροπή σας και η Κομισιόν για σύστημα αξιολόγησης. Οπότε έτσι έχουμε ένα ολόκληρο θεματολόγιο με το οποίο θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τα πράγματα τα μέσα επόμενα χρόνια. Δεύτερο η κυρία Κέρτον Γκάλαντ. Σας ευχαριστώ και πάλι. Και ε, μας αναφέρετε ένα σωρό ζητήματα. Εμεί όμω την τελευταία πενταετία αυτό το οποίο είδαμε είναι ότι Υπάρχει το καρότο, αλλά σπάνια εμφανίζεται το μπαστούνι σε σχέση με ε, το θέμα αυτό της γενικευμένες προτιμήσεις. Ναι, αλλά στη συνέχεια της πρώτης τι θα γίνει με τις υποχρεώσεις των ε, επενδυτών. Όλα λέμε για τα δικαιώματά τους, ε, το ISDS που θα μεταμορφωθεί. Όμως θα κάνετε τίποτα για αυτό το καυτό θέμα και τις υποχρεώσεις του επενδυτού. Και έτσι οι ευρωπαϊκές ε, ε, επιχειρήσεις που επενδύουν στον κόσμο να σέβονται τα ανθρωπινά δικαιώματα και γενικά σύνομα να ακολουθούν όλη την αλυσίδα της προσφοράς. Γίνεται αυτό, λέει ο με τα προγράμματα που αφορούν την Τράπεζα Επενδύσεων και άλλα προγράμματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όταν ήμουν επιτροπό Γεωργία, είχα εξοικειωθεί πολύ με το θέμα. Να, στην Αφρική. Στην Αφρική πολλές φορές μας επέκραναν γιατί δεν κάνουμε περισσότερα για να εξασφαλιστεί ότι θα υπάρχουν υπεύθυνε επενδύσεις. Οπότε και εμεί σε συνεννόηση με την Αφρικανική Ένωση καταλήξαμε σε συμφωνία. Ο καθένα τώρα ξέρει το ρόλο του, πολιτική αποφασιστικότητα, χρηματοοικονομική υποστήριξη. Έτσι είμαστε πιο υπεύθυνοι. Ένα σωρό προγράμματα υπάρχουν. Αλλά βέβαια και οι ιδιώτες θα πρέπει να φέρονται υπεύθυνα και αυτό που θα δούμε να πετύχουμε και προς εκείνη την κατεύθυνση. Ούτως ώστε να τηρούν τις υποχρεώσεις τους οι επενδυτές. Ο πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριος Μπιουτικόφερ. Καλησπέρα. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι το οποίο έθιξε η κυρία Φανμπρέμπτ. Το κατεπήγον της κλιματικής κρίσης σημαίνει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και τις εμπορικές συμφωνίες. Το μόνο το οποίο λέτε στην επιστολή σας είναι ότι θα υπάρξει κεφάλαιο βιώσιμης ανάπτυξης Τελεία και παύλα. Μάπα το καρπούζι. Ε, λέτε ότι ε, θεωρείτε ότι είναι σημαντικά αυτά τα κεφάλαια. Ε, επιδείξτε λίγη φιλοδοξία, σας παρακαλώ. Είναι επαρκείς ως έχουν. Πώς προτείνετε να ενισχυθούν. Τι είστε διατεθειμένος να κάνετε έτσι ώστε να είναι εφαρμόσιμες και να μπορούν να επιβληθούν οι περιβαλλοντικές προδιαγραφές συμφωνίας ελευθεροπορίου. Απάντηση. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα οι διεθνείς ε, συμφωνίες μας ε, να ενσωματώνονται σε εμπορικές συμφωνίες και ε, να μπορούν να επιβληθούν σε διμερές, πολυμερές επίπεδο. Τώρα δεν είμαι σίγουρος το ποιες ε, χώρες εννοείται σε σχέση με τις συμβάσεις για τα εργασιακά, γιατί έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ακόμα και με το Βιετνάμ, όπου ε, σημειώνουμε σημαντική πρόοδο με τις 8 συμβάσεις και πριν από την κύρωση της ε, συμφωνίας για να επηρεαστούν, για να, με συγχωρείτε, για να κυρωθούν κάποιες από αυτές τις συμφωνίες. Και Παραγουάι, και Αργεντίνα έχουν κυρώσει και εφαρμόσει όλες της ε, συμφωνία για τα Εργασιακά. Μία έχει απομείνει στη Βραζιλία. Αλλά η δικιά μου φιλοδοξία είναι να ενσωματωθούν αυτά στο μέτρο του δυνατού και με όσο το δυνατόν ε, περισσότερη πολιτική πίεση και με την έγκριση του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σας οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε μιλάμε για οικονομικές είτε περιβαλλοντικές και κοινωνικές. Κύριε Επίτροπε, αναφέρατε μόλις την Κίνα και διαβάζω εδώ πέρα πως ε, σκοπεύετε να επιτύχετε μια συμφωνία μέχρι το 2020. Αυτό σημαίνει ότι θα οριστικοποιηθεί η συμφωνία ε, υπό οποιασδήποτε συνθήκε Σημασία έχει η ουσία, όχι η ταχύτητα. Το δικό μου το ερώτημα για τον αρμόδιο για την επιβολή των συμφωνιών είναι το εξής. Μπορείτε να δεσμευτείτε ότι αυτός ο αρμόδιος ε, θα διαβουλεύεται τακτικά, όχι μόνο με τις επιχειρήσεις, αλλά και με τα συνδικάτα και την κοινωνία των πολιτών και η αρμόδια αυτή θα μπορεί να ασχολείται με καταγγελίες αυτών των ενδιαφερομένων. Θα σας δώσω οποιαδήποτε διαβεβαίωση θέλετε για όσο δυνατόν περισσότερες επαφές το εμπόριο είναι πολύ σημαντικό οικονομικό μέσο, αλλά βεβαίω ε, αγγίζει και πολλές άλλες περιβαλλοντικές πτυχές που θέλουμε να ενσωματώσουμε στις ε, συμφωνίες αυτές ε, στο πλαίσιο της πολιτικής περί δημοσίων αγαθών, τις οποίες γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Οπότε έχετε την δέσμευσή μου ότι θα διαβουλευτούμε με όλους τους ενδιαφερόμενους και οπωσδήποτε το Κοινοβούλιο, την Επιτροπή σας. Εγώ θα είμαι σε επαφή με όλους και θα έχουμε έναν ρόλο γενικό για την εφαρμογή. Δεν θα κάνω καμία δέσμευση τώρα για ε, καταγγελίες. Δεν θέλω να γίνω ε, ένας ακόμα διαμεσολαβητής. Θέλω να δω τι δομή θα έχουν όλα αυτά, γιατί δεν θα έχουμε τους ίδιους πόρους ε, για να υποκαταστήσουμε τον διαμεσολαβητή. Αλλά είμαι διατεθειμένος να συζητήσω αυτά τα οποία θέλετε για να εστιάσουμε στις καταγγελίες γιατί όπως έχουμε και με το παράδειγμα του Περού ε, έχουμε εστιάσει στην κοινωνία των πολιτών και τελικά καταλήξαμε σε ένα σχέδιο δράση για να εφαρμόσουμε το σχετικό κεφάλαιο. Οπότε μια τέτοια ε, διαδικασία θα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δούμε τώρα. Αλλά χωρίς να κάνουμε δύο φορές την ίδια δουλειά, έτσι, με άλλες υπηρεσίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Ραφαέλα έχει τον λόγο. Τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση συνήψε Συμφωνία στις οικονομικές εταιρικέ σχέσει με αφρικανικές περιοχές και χώρες. Δύο περιφερειακές και διαφορετικού λόγους να σταματήσει. Ανατολική και Δυτική Αφρική. Θα επικαιροποιηθεί αυτή η συμφωνία σε μια ευρύτερη συμφωνία που θα περιλαμβάνει πρότυπα αηφορία. Πώ θα εξασφαλίσετε ότι η συμφωνία μετά το κοτονί, μάλλον οι εμπορικέ σχέσει μετά το κοτονού μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Αφρική θα βασίζονται σε αξίε, θα συνάδουν με το θεματολόγιο τη Ένωση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και θα χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη ισότητα. Θα πρέπει λοιπόν να αναβαθμιστεί η Συμφωνία Εταιρική Σχέση για να λαμβάνει υπόψη και κριτήρια βιωσιμότητα και ισότητα των φύλων. Και επίση, τι θα πει μεγαλύτερη ισότητα σε αυτό το πλαίσιο, κατά την άποψή σα πάντα. Απάντηση. Όπως γνωρίζετε, η υποψήφια πρόεδρος της Κομισιόν ζήτησε μια πλήρη συνεκτική στρατηγική για την Αφρική, όπου θα περιλαμβάνονται και στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης εκφύσεως δηλαδή, θα βασίζονται σε αξίες και θα περιλαμβάνεται και το ζήτημα του φύλου. Ήδη έχω εργαστεί στο πλαίσιο TPS και για να στηρίξουν εφαρμογή των συμφωνιών με τις χώρες αφρικανικές. Παρήχαμε και τεχνική βοήθεια. Η κυρία Σάκο ήταν ε, η αρμόδια. Μετά το Κοτονού τώρα. Έχουμε διαβουλεύσει, αναφέρεται για να ενισχύσουμε την εταιρική σχέση με την Αφρική προς την ίδια κατεύθυνση. Θέλουμε βιώσιμη ανάπτυξη και κοινέ αξίες. Ανατολική Αφρική τώρα. Πράγματι, ε, αργά κινούνται αλλά νομίζω ότι αύριο ξημερώνει μια νέα μέρα σε ό,τι αφορά τη σχέση μας με την Ανατολική Αφρική και την ανάπτυξη μιας νέας συμφωνίας ε, εταιρική σχέση που θα μπορούσε ενδεχομένω να αναβαθμιστεί σε εμπορική συμφωνία, σε συμφωνία ελεύθερου εμπορίου. Γιατί η EPA μέχρι στιγμή δεν περιλαμβάνει αυτά, δηλαδή η συμφωνία οικονομική εταιρική ε, σχέση. Και αν μπορώ να κάνω οτιδήποτε για να βοηθήσω να έχουμε συμπερίληψη όλων αυτών, θα το κάνω. Επερώτηση για το εμπόριο και το φύλλο. Εμβαθύνω λίγο σε αυτό. Είναι επιτυχημένη αυτή η προσέγγιση να χρησιμοποιούμε το εμπόριο για άλλους στόχους. Άρα θα έπρεπε να είναι ε, η διάσταση του φύλου μεταξύ αυτών των στόχων η ε, Μάλστρομ ε, στην εντολή τη έλαβε πολύ σοβαρή υπόψη τη διάσταση του φύλου και σε μία διάσκεψη σήμερα επί Τι θα κάνετε εσεί στο πλαίσιο του διεθνού εμπορίου, ώστε οικονομικά, οικονομική, κοινωνική θέση και δικαιώματα να γίνονται σεβαστά. Θα ε, ακολουθήσετε τα βήματα τη κυρία Μάλστρομ, ώστε να υπάρχουν διατάξει ε, που θα αναφέρονται στο φύλλο στι μελλοντικέ συμφωνίε. Αυτό είναι ναι ή όχι. Θα είναι ένα ναι ή ένα όχι. Πράγματι ήταν μεγάλη επιτυχία της κυρίας Μανστρόμ τα περί ισότητας των φύλων. Σε μια από τις γραπτές μου απαντήσεις είπα ότι σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της πολιτικής μου θα δώσω εντολή στις υπηρεσίες μου να λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο του φύλου στις πρωτοβουλίες της πολιτικές ε, που θα προωθήσουμε στο μέλλον. Ξέρω ότι η κυρία Μάλστρομ είχε πολύ επιτυχημένη διάσκεψη σήμερα. Με ενημέρωσαν από αυτού. Και σήμερα είπε και η ίδια και ο Γενικός Διευθυντής ότι υπάρχει και έντονο οικονομικό σκεπτικό ε, πίσω από αυτό. Τη συμπερίψη του φίλου. 28-3 δολάρια θα μπορούσαν μέχρι το 2025 να είναι το κέρδος από τη χειραφή των γυναικών. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικά τα ε, διακυβευόμενα και θα το έχουμε υπόψη μα και για τι διαπραγματεύσει μα στο πλαίσιο συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου το θέμα τη διάσταση του φύλου. Ο Γιούλιο Βίνκλερ είναι ο τελευταίο ομιλητή. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ υποψήφιε επίτροπε. Δεν ξέρω αν κάνω λάθο, αλλά έχω την εντύπωση ότι ο ελέφαντα σε αυτό το Mission Letter είναι η Κίνα και άλλου ελέφαντε συζητήσαμε. Σήμερα η Κίνα όμω είναι ο ελέφαντα με ε κεφαλαίο στην αποστολή σας όπως την αναφέρει η κυρία Φοντερ Λάιεν και αν δεν υπάρχει ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού, ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ανησυχούν μας, το λένε ξεκάθαρα, υπάρχει στρέβλος της αγοράς και από την άλλη πλευρά θέλουμε να βελτιώσουμε και τις προοπτικές της συνολικής συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας. Θέλουμε να συμφωνήσουμε τι γεωγραφικέ συνδείξεις και πολλά άλλα. Αλλά υπάρχει μια αντίφαση. Όλα αυτά τα θέματα είναι επίμαχα και η δική σας προσέγγιση ποια θα είναι. Γιατί πρόκειται για δύσκολα θέματα. Και εταίροι σα ε, για την προσέγγιση με την Κίνα, ποιοι θα είναι ε, από την, από την έκομψη. Κύριος Κογκο, όλοι. Και η πρόεδρος και όλοι οι επίτροποι. Αλλά κυρίως αντιπρόεδρος ε, ε, Βάλτης Ντομπρόσκης για την οικονομική ανάπτυξη. Θα έχω στενή σχέση με αυτόν, αλλά και για τα θέματα της περιβαλλοντικής αηφορίας, κλιματικής αλλαγής, ε, με τον αντιπρόεδρο Τίμερμανς. Και βέβαια, όπως ξέρετε, υποχρεούμε και με τον αντιπρόεδρο Βεστάγκερ για το ψυχιακό εμπόριο να έχω ε, πολύ στενή συνεργασία. Με όλους θα συζητήσω και η κυρία Φοντρελάιν είμαι σίγουρο, ότι θα στρέφεται συχνά στο θέμα αυτό και θα με ρωτάει. Γιατί έχει βάλει πολύ φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα τα τέλη του 2020. Έχω ξεκινήσει 5 Νοεμβρίου. Πρώτη μου επίσκεψη εκτός Ευρώπης στην Κίνα και η Υπουργική Διάσκεψη του ΠΟΕ. Ελπίζω εκεί να μπορέσω να ε, έχω επαφές με τους Κινέζους κάθε πέντε χρόνια αλλάζει η Κομισιόν, είναι ευκαιρία να ξαναορίσουμε τις προτεραιότητές μας και το θεματολογιό μας. Νομίζω θα συνεχίσουμε την στρατηγική για την Κίνα, δηλαδή έχουμε εργαλεία στη διάθεσή μας και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των αθέμητων εμπορικών πρακτικών. Θέλουμε να έχουμε στο δυνατόν πιο ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού. Ταυτόχρονα υπάρχουν και πολλά που πρέπει να γίνουν. Όταν λένε οι Κινέζοι ότι θα ανοίξουν την αγορά τους, πρέπει να το κάνουν στην πράξη και δεν το έχουν κάνει μέχρι τώρα. Μέσω της επενδυτικής συμφωνίας θα δούμε αν μπορέσουμε να έχουμε στόχους ε, και κάποιους ε, ε, σταθμούς που θα πρέπει να... Γιατί δεν μπορεί να είναι οι μόνοι ωφελημένοι για, από τη συμμετοχή τους στον ΠΟΕ οι Κινέζοι ε, έχουν σίγουρα κερδίσει πολλά, αλλά πρέπει να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις τους. Και αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε ως μόχλευση. Γιατί υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα μέχρι το 2020 που πρέπει να κλείσουν. Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Και επειδή έχω το προνόμιο να είμαι ο τελευταίος που κάνει ερωτήσεις ε, από την Επιτροπή μας, μια ερώτηση για τη Γεωργία. Γιατί πολλοί συνάδελφοι αναφέρονται στη Γεωργία. Είναι σημαντικά πολλά θέματα, παράδειγμα χάρη. Συνεργασία και η σχέση εμπορίου και γεωργίας είναι σημαντική και είναι κάτι που σας ενδιαφέρει, είναι προσφυλές στο θέμα της γεωργίας, είναι και το χαρτοφυλακιό σας, αλλά πρέπει να δούμε τις προκλήσεις για τους αγρότες, ε, που είναι αυτά που περιλαμβάνουν οι συμφωνίες ελεύθερου. Αλλά δεν είναι μόνο προκλήσεις, μιλάμε και για πολλές ευκαιρίες για τους γεωργούς, ε, για την αγρομηχανία. Ε, και η ερώτησή μου είναι τι θα κάνετε επίτροπε ω αρμόδιο πλέον για το εμπόριο Επίτροπο, για να βοηθήσετε τους αγρότες να εκμεταλλευτούν περισσότερο τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου της Ένωσης απάντηση. Όπως γνωρίζετε κύριε Βίνκλερ, οι αγρότες δεν σας λένε τα καλά νέα για τις ε, συμφωνίες. Ποτέ δεν λένε μια καλή, κάτι, κάτι καλό, κάποιο καλό. Και πάντα προσπαθούν να, ε, να τα κρατάνε αυτά μυστικά, καλά κρυμμένα. Τα ξέρω κι εγώ σαν αγρότες. Με την Ιαπωνία. Έχουμε ίσω τη μεγαλύτερη και πιο φιλόδοξη, ιδίως τα τη Γεωργία, εμπορική συμφωνία. Έχουμε 98% απελευθέρωση. Τεράστιες επίσης ε, ευκαιρίες με τον Καναδά έχουμε, με το Μεξικό. Υπάρχουν πολλές περιοχές. Και ανάλογα με τα ισχυρά σημεία ή το ε, ενδιαφέρον που έχουν οι διάφορες χώρες, θα εστιάζουν κάπως συγκεκριμένα. Έχουμε πάρα πολλές θέσεις εργασίας για την Ήπεθρο, για τις αγροτικές περιοχές. Έχουμε λοιπόν ένα συμφέρον ε, να φροντίσουμε να εφαρμόζονται εμπορικές συμφωνίες, οικονομικό, περιβαλλοντικό, κοινωνικό συμφέρον, φυσικά στη Γεωργία. Ε, υπάρχουν και 200 εκατομμύρια για το γεωργοδιατροφικό κλάδο που τα, που τα βάζουμε το 2020 για την προώθηση κλάδου. Είχαμε το 2015 την κρίση στον ε, κομικό τομέα και εγώ έκανα πολλές αποστολές, 20 ε, τουλάχιστον. Θέλαμε να βοηθήσουμε ε, να αυξηθούν οι πωλήσει των υψηλή ποιότητα ευρωπαϊκών προϊόντων. Και αν θέλετε να σα πω κάτι, η ποιότητα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αν μειωθεί η ποιότητα, και η μεσαία τάξη θα συρρυκνωθεί, ιδίω στην Ασία. Γιατί θέλουν. Η βιωσιμότητα είναι κάτι πολύ σημαντικό στην παραγωγή, στην μεταποίηση. Αυτό θέλει η αγορά. Κοντόθωρο θα ήταν ε, από το διατροφικό κλάδο και τους αγρότες μας να μην επενδύσουν ε, στην ε, βιωσιμότητα και στην ποιότητα των προϊόντων. Ως αρμόδιος για το εμπόριο επίτροπος ελπίζω να έχω έναν επίτροπο αρμόδιο για τη Γεωργία με τον οποίο θα μπορώ να συνεργάζομαι με ολοκληρωμένο τρόπο για να βελτιστοποιήσουμε και να μεγιστοποιήσουμε την εφαρμογή των συμφωνιών προς όφελος και των αγροτών. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ υποψήφιε επίτροπε για τις απαντήσεις. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους για τις ερωτήσεις. Είναι σαφές λοιπόν πως ε, εδώ πέρα είναι η καρδιά της δημοκρατίας όσον αφορά την εμπορική πολιτική και όλα τα επίμαχα θέματα νομίζω έχουν καλυφθεί και έχει άρα ξεκαθαρίσει το ότι ο καιρός που οι πολιτικοί χαράζονταν πίσω από κλειστές πόρτες έχει παρέλθει και χρειάζεται διαφάνεια στην διαμόρφωσή της. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, έχετε τώρα την δυνατότητα να συνοψίσετε την συζήτηση και να κάνετε κάποιες παρατηρήσεις. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ που είχατε την ευγένεια να με δεχτείτε απόψε και ευχαριστώ και για τις κέρυες ερωτήσεις σας. Ελπίζω να απάντησα στο μέτρο των ικανοτήτων μου. Ίσως ε, θεωρείτε ότι ήταν κάπως ε, σύντομες γιατί σε 15 μέρες ε, προσπάθησα να εμβαθύνω στα ζητήματα αυτά αλλά υπόσχομαι να επανορθώσω εάν με εγκρίνεται. Αλλά θεωρώ ότι το εμπόριο είναι σημαντικό, είναι κάτι το βασικό για τα ανθρώπινα όντα το εμπόριο από την εποχή του λίθου. Έχουν βρεθεί στοιχεία ότι πριν ε, ε, καταλήξουν οι κυνηγοί τροφοσυλλέκτες να γίνουν γεωργοί, αντάλλασαν ε, διάφορα αντικείμενα μεταξύ τους. Οπότε είναι θέμα και περηφάνειας αισιοδοξία, εξερεύνησης και βεβαίως καινοτομίας και κινδύνου και κυρίως είναι ένα ζήτημα εμπιστοσύνης. Και βεβαίως όταν πιάνουμε ένα στυλό και υπογράφουμε και λέμε αυτοί είναι οι κανόνες και αυτές είναι οι μέθοδοι συμμόρφωσης, ε, αυτή είναι η εμπιστοσύνη. Και έτσι έχει ακριβώς οικοδομή στην φήμη της η Ευρωπαϊκή Ένωση ως αξιόπιστος και έμπιστος εταίρος, γιατί εμείς πάντα θεωρούμε ότι είμαστε εταίροι και τα πράγματα είναι σαφή και στις δύο πλευρές. Και πριν ε, γίνει της μόδας ε, το περιβάλλον, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη είχε ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα και ξεκινούσαμε από την παραγωγή, από τους σπόρους ε, που φυτεύαμε και ακριβώς ε, θέλουμε η παραγωγή μας να βασίζεται στην αηφορία. Λοιπόν το εμπόριο και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως στόχο το να ωφελούνται όλοι, όχι μόνο μερικοί και το ίδιο αισθάνονται και όλα τα κράτη-μέλη και όλοι οι γεωργοί και ε, εξ ανάγκης βεβαίως πρέπει η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να χαράστε σε πολύ μεγάλο επίπεδο. Ποτέ δεν πρέπει να ξεχνά το άτομο. Το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, κύριε Πρόεδρε, ξεκίνησε από το χάος και την καταστροφή μέσα στα συντρίμια. Οι Ευρωπαίοι φαντάστηκαν κάτι καλύτερο και ξεκίνησαν να το οικοδομούν. Ε, έθεσαν ε, αδύνατους στόχους και πολλές φορές τα κατάφεραν και μέσω του εμπορίου. Ναι, βεβαίω, ε, η νομοθεσία και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχουν σημαντικό ρόλο, αλλά το εμπόριο έχει παίξει εξίσου σημαντικό ρόλο και ίσως να παίξει και ακόμα σημαντικότερο στο μέλλον. Έχει σημασία λοιπόν το πώ εμπορευόμαστε. Το πώ εμπορευόμαστε δείχνει το ποιοι είμαστε και το τι αξίες έχουμε. Έχει έναν τεράστιο αντίκτυπο στον υπόλοιπο κόσμο, όπως ξέρουμε και από τη συζήτηση που ακούσαμε απόψε. Οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι ένα ισχυρό παγκόσμιο παίκτη και να παίξει ηγετικό ρόλο στο εμπόριο. Κάθε πτυχή τη εμπορική πολιτική θα πρέπει να επιδεικνύει τοπικά και παγκοσμίω την δεσμευσή μα στην ειρήνη, την ευημερία και στο να σταματήσουμε την περιβαλλοντική ρήπανση. Αυτό πιστεύω και ελπίζω ε, να ε, έχω την εμπιστοσύνη σας ως Επιτροπός για το θέμα αυτό για να το αποδείξω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thanks lot, Commissioner Ευχαριστούμε πολύ κύριε υποψήφιε Επίτροπε, λέει ο Και τώρα είναι η σειρά των πολιτικών ομάδων. Γιατί σε μισή ώρα τώρα μέχρι τις ε, και μισή και κλεισμένων θα συζητήσουν και θα συζητήσουμε εδώ για την ετοιμιγορία μας σχετικά με την ακρόαση. Σας ευχαριστώ πολύ.